Αγαπητοί συνάδελφοι, χαρά μου που σας καλωσορίζω στην ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής μας, την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν για τυπικούς λόγους να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Έχετε παρατηρήσει στην ημερήσια διάταξη, όχι. Ωραία, εγκρίνεται. Οπότε περνάμε απευθεία στο κύριο θέμα της έκτακτη συνεδρίασής μας και καλωσορίζω θερμά τον πρόεδρο του Eurogroup, τον Χερούν Ντάιζελμπλουμ, για την τακτική ε, συζήτηση για τα οικονομικά θέματα σύμφωνα με τους κανόνες, με το άρθρο 2b του κανονισμού του 1997-466 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό 1175 του 2011. Αυτές οι τακτικές συναντήσεις ε, θέλω λοιπόν να επενθυμίσω ότι ε, γίνονται με ε, με νομική βάση. Έχουμε αυτήν την ε, εξαμηνιαία συνάντηση διαλόγου με τον πρόεδρο του Eurogroup. Είναι τώρα λοιπόν η αρεινή και θα έχουμε και φθινοπορεινή συνάντηση. Η τελευταία έγινε στις 29 Δεκάτου παρελθόντος έτους. Στην εδρία λοιπόν σήμερα ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το πρόγραμμα εργασιών του Eurogroup για το πρώτο εξάμεινο του 2017 το Eurogroup εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών κάθε εξάμεινο που καθορίζει διάφορους ε, τομεί όπου πρόκειται να εστιάσει τι προσπάθειέ του το Eurogroup. Η Επιτροπή μου θα ήθελε επίσης, η Επιτροπή μας θα αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να ακούσει και για τα πορίσματα της ε, χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup. Ιδιαίτερα δύο θέματα που ήταν στην ημερήσια διάταξη, αποτίμηση του Eurogroup για την πρόοδο, για τη δεύτερη αξιολόγηση του μακροοικονομικού προγράμματο στην Ελλάδα και δεύτερον, η συνέχιση της εφαρμογής του, των σχεδίων ε, δημοσιονομικού προγραμματισμού για το 2017 και της δημοσιονομικής κατάστασης στην ε, Ευρωζώνη. Σύμφωνα με το 2PAC, ε, τα, το σχέδιο δημοσιονομικών προγραμμάτων θα εξεταστεί πριν από την τελική έγκρισή του από το ΕΚΟΦΗΝ. Ξέρετε τους κανόνες. Θα ξεκινήσουμε με την ε, εισαγωγική δήλωση του Προέδρου του Eurogroup και μετά θα έχουμε ερωταπαντήσεις με τα μέλη της Επιτροπής μας. Πέντε λεπτά, ως συνήθως. Λοιπόν, για να μην καθυστερήσουμε, όλοι ξέρετε πολύ καλά τη διαδικασία, να δώσω λοιπόν με χαρά το λόγο στον Χερούν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πάρω το λόγο ενώπιόν σας και μαζί σας για άλλη μια φορά στις τακτικές αυτές συναντήσεις που έχουμε. Καταρχάς θα ήθελα να επικεντρωθώ στις οικονομικές προοπτικές και στη συνέχεια θα μιλήσω για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό για την εργασία του Eurogroup. Καταρχάς να ξεκινήσω τονίζοντας ότι έχουμε ορισμένες θετικές εξελίξεις ο πρόσφατος γύρος προβλέψεων από διεθνείς οργανισμούς επιβεβαίωσε ότι η Ευρωζώνη εισέρχεται στο τέταρτο συναπτό έτος οικονομικής ανάκαμψης και η θετική οικονομική ανάκαμψη προβλέπεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Έχουμε όμως και άλλα θετικά σημάδια στην αγορά εργασία, για παράδειγμα. Το ποσοστό ανεργία στην Ευρωζώνη να μένεται να συνεχίσει τη σταθερή πτωτική του τάση όπως όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τη Eurostat βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από το 2009. Αλλά είναι ακόμα βέβαια αρκετά υψηλό, πολύ υψηλό αυτό το ποσοστό. Είναι θερετική πάντως η πτωτική αυτή στάση, ιδίως επειδή βλέπουμε ότι η ανάπτυξη έχει διαρκώς πιο ευρία βάση με αξιοπρεπή ποσοστά μεγέθυνση και βελτιωμένα δεδομένα για την απασχόληση παντού στην Ευρωζώνη. Οι δημοσιονομικέ και άλλε μακροοικονομικέ ανισορροπίε συνεχίζουν να υποχωρούν. Έχουμε δει αρκετέ σημαντικέ μετατροπέ του 2016, ωστόσο η Ευρωζώνη όμω παρέμεινε ανθεκτική, μόνο ότι υπάρχει αβεβαιότητα που επικρατεί βέβαια σε πολλά μέτωπα. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια σαφή ένδειξη ότι οι αναγκαίε και μερικέ φορέ δύσκολε μεταρρυθμίσει που εφαρμόζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αποδίδουν καρπού. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι, παρόλα αυτά όμω δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Παρά τι σαφεί βελτιώσει που βλέπουμε, τα κληροδοτήματα τη κρίση εξακολουθούν να ανακόπτουν μια δυνάμει ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη. Και έτσι περνάω στο θεματολόγιο πολιτική που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Η διασφάλιση μια ανάπτυξη χωρί αποκλεισμού. Αυτό θα πρέπει να είναι η πρωταρχική μα προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να δημιουργήσει ακόμα περισσότερε θέσει εργασία και όπου κρίνεται αναγκαίο συμμετοχή στην αγορά εργασία όσων έχουν ήδη μία δουλειά θα πρέπει να αυξηθεί. Πρέπει να διασφαλίσουμε επίση την ανταγωνιστικότητά μα, αλλά παράλληλα θα πρέπει να έχουμε κέρδη παραγωγικότητα και όχι μόνο συγκράτηση του κόστου. Μολονότι οι προτεραιότητε διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, η απάντηση στι προκλήσει αυτέ είναι κοινή για όλου. Εξαρτάται πρωτίστως, από την αποφασιστική εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να απελευθερωθεί η παραγωγική ικανότητα που αναμφίβολα διαθέτει η Ευρωζώνη. Οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει καθιστούν τι αγορέ εργασία και τι αγορέ προϊόντων μα πιο σύγχρονε, πιο φιλικέ για τι επιχειρήσει και πιο αποτελεσματικέ. Θα πρέπει όμω να συνεχίσουμε και με τη στρατηγική διόρθωση των ισολογισμών, προκειμένου να διορθώσουμε το υπερβολικό χρέο του ιδιωτικού τομέα. Χρειάζονται λοιπόν πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά ρυθμιστικά πλαίσια για την αφαιρεγκαιότητα με τη μέγιστη δυνατή εναρμόνιση. Η πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκθέσεις αναχώρα λέει ότι έχει γίνει περιορισμένη πρόοδος στην εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα. Η περιορισμένη λοιπόν αυτή πρόοδος για τις δραστικές μεταρρυθμίσεις είναι λυπηρή. Και τονίζω, ουσιαστικά ότι θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε το συντονισμό της πολιτικής μας με μια βαθμία μετάβαση σε ένα σύστημα συγκρατικής αξιολόγησης. Το Eurogroup διερευνά αυτή τη δυνατότητα σε διάφορου τομεί στο πλαίσιο των θεματικών συζητήσεων που κάνουμε για την ανάπτυξη και τι θέσει απασχόληση. Εμεί συζητήσαμε το ζήτημα τη συγκριτική αξιολόγηση στα πλαίσια τη βιωσιμότητα του στεξιωτικού συστήματο στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup. Α περάσω τώρα στο ρόλο τη δημοσιονομική πολιτική. Το Eurogroup συζήτησε το ζήτημα του κατάλληλου δημοσιονομικού προσανατολισμού στην Ευρωζώνη Πολλέ φορές στο παρελθόν, πιο πρόσφατα το Δεκέμβριο, όταν συζητήσαμε τα σχέδια προπολογισμού, τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των, των κρατών μελών της Ευρωζώνης για το 2017. Η γενικότερη συνένεση είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην χρησιμοποίηση του δημοσιονομικού χώρου για την ενίσχυση της οικονομίας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών. Βλέπουμε όμως ότι τα ποσοστά δημόσιου χρέους είναι ιδιαίτερα υψηλά και υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο για να κάνουμε τη διάρθρωση των εθνικών προπολογισμών πιο φιλική προς την ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να συμμορφούνται πλήρως τα κράτη-μέλη με, με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και να συμμορφώνται με τους κανόνες που βλέπουμε στο σύμφωνο αυτό. Εμείς θα παρακολουθούμε εκ του σύνογγι στην δημοσιονομική αυτή κατάσταση. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό στη συνεδρίαση του Μαΐου, έχοντας υπόψη μας τις αρινές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα δούμε τότε πώς εφαρμόζονται αυτά τα σχέδια προπολογισμού και ποιες είναι οι αλλαγές που έχουν λάβει η χώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίζονται, να συμμορφούνται τα κράτη-μέλη με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το οποίο θα αναθεωρήσουμε εν ευθέτω χρόνο. Θα ήθελα να περάσω τώρα στο πρόγραμμα για την Ελλάδα. Όπω ξέρετε, οι ελληνικέ αρχέ συνεργάζονται με του θεσμού και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για μια πλήρη δέσμη μεταρρυθμίσεων. Ήδη τον προηγούμενο μήνα στο Eurogroup κατέληξαν σε μια κοινή αντίληψη ότι η δέσμη αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει εκ των προτέρων διαρθρωτικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν κάποια στιγμή λίγο αργότερα, προκειμένου να γίνει πιο εύρωστη η οικονομία της Ελλάδας και πιο φιλική προς την ανάπτυξη και ότι θα πρέπει να έχουμε και τα απαραίτητα επεκτατικά δημοσιονομικά μέτρα προκειμένου να καλύψουμε πιθανή υπερκάλυψη των δημοσιονομικών στόχων. Είναι πολύ σημαντική μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και αυτό αποτελεί σημαντικό τμήμα των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να εξορροπηθεί ο εξυγχρονισμό τη οικονομία με τον αγκαίο σεβασμό για τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων σύμφωνα με τι ευρωπαϊκέ βέλτιστε πρακτικέ. Παράλληλα, οι εταίροι τη Ελλάδα στην Ευρωζώνη τήρησαν τη δέσμευση που ανέλαβαν το Μάιο του 2016 και ενέκριναν μια δέσμη βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέο για να μειώσουν τον κίνδυνο επιτοκίου σχετικά με το δημόσιο χρέο τη Ελλάδα. Και η εφαρμογή βέβαια των μέτρων αυτών είναι εν εξελίξη. Τώρα, τις επόμενες ημέρες συμφωνήσαμε ήδη χθε ότι θα εντατικοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις και συζητήσεις μεταξύ των θεσμών και των ελληνικών αρχών εδώ στις Βρυξέλλες, προκειμένου να ασχοληθούμε με τα πιο βασικά εκκρεμή ζητήματα προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε μια συμφωνία σε αυτά και στη συνέχεια θα οριστικοποιήσουμε όλα τα υπόλοιπα εκρεμή ζητήματα προκειμένου να καταφέρουμε να συζητήσουμε αυτά στα πλαίσια του Eurogroup και προκειμένου να κάνουμε εκεί πέρα μια πιο πολιτική συζήτηση. Και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει τον Απρίλιο και αν όχι τον Απρίλιο, τον Μάιο. Αυτή είναι η βασική φιλοδοξία επί της οποίας συμφωνήσαμε χθες και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές τις συνομιλίες. Ολοκληρώνω σε αυτό το σημείο κύριε Πρόεδρε και αφήνω κατά αυτόν τον τρόπο χρόνο για ερωτήσει. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτήν την ε, σύντομη εισαγωγή η οποία δίνει και αρκετό χρόνο στους συναδέλφους για να πάρουν το λόγο. Ξεκινάμε λοιπόν. Κατ' από την ε, πλευρά του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και ευχαριστούμε τον πρόεδρο Ντάσιμπλουμ. Καταρχήν, Ελπίζουμε να είναι ενδιαφέρουσα η σημερινή συζήτηση που κάνουμε αφού ολοκληρώθηκε και η προεκλογική εκστρατεία στη χώρα σας. Και από την πλευρά μου θα ήθελα να θέσω δύο ζητήματα προς συζήτηση. Το ένα είναι η λευκή βίβλος σε ό,τι αφορά το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη και την 20η επέτειο από την υπογραφή των συνθηκών της, της δρόμης ε, και λαμβάνοντα υπόψη και τη σχετική ανακοίνωση τη Επιτροπή, ε, διαρχόμαστε μία περίοδο αναλογισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακριβώ με βάση αυτό το υπόβαθρο θα ήταν από του Προέδρου του Eurogroup πώ θα συμβάλλει το Eurogroup σε αυτή τη διαδικασία ακριβώ και στο πλαίσιο του ε, της μελλοντικής διαμόρφωσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα ε, ποιες μεταρρυθμίσεις θεωρείτε πως είναι οι πλέον επίγουσες σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και επίσης γνωρίζουμε ότι θέλετε να υπάρχει μια μόνιμη προεδρία του Eurogroup Κροβάλλου εκεί και μετά έχετε άλλες προτάσεις για το μέλλον της Ένωσης αυτής. Θα περιοριστώ μόνο σε αυτά τα ερωτήματα για να σας δώσω τη δυνατότητα να τα απαντήσετε, να τεθούν και περαιτέρω ερωτήματα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βάση για αυτά τα ερωτήματα. λευκή βίβλος της Επιτροπής θεωρώ πως ε, είχε νόημα γιατί πραγματικά περιέγραφε μία σειρά από σενάρια, τα οποία καταδεικνύουν τελικά ποιε είναι εναλλακτικέ που έχουμε μπροστά μα. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα συνδυασμού κάποιων από αυτά τα σενάρια. Δηλαδή, ε, μπορεί να υπάρξει το σενάριο όπου κάποια μικρά κρατημέλη αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο σε ε, κάποια ζητήματα επιτρέποντα την εστίαση των προσπαθειών που γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση σε ορισμένα σταδιακή σημασία ζητήματα και όπου είναι ε, ξεκάθαρη η προστιθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντα κατά μέρο άλλα ζητήματα των οποίων μπορούν να επιλεφθούν οι εθνικέ ε, κυβερνήσει. Άρα λοιπόν θεωρώ πω πραγματικά προσεγγίζει με σωστό τρόπο αυτή η λευκή δήλωση τη Επιτροπή το ζήτημα και υπενθυμίζω ότι μπορούμε να συνδυάσουμε κάποια από τα σενάρια που περιλαμβάνει. Ε, το Μάιο θα υπάρξει ένα έγγραφο από την πλευρά μα σε ό,τι αφορά το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, το οποίο προφανώς θα συζητηθεί στο Eurogroup, αλλά θα πρέπει να συζητηθεί και σε επίπεδο Συμβουλίου Αγκοφήν. Και αυτό γιατί προφανώς και τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ ενδιαφέρονται ακριβώς ε, και θέλουν να παραμείνουν μέσα στην όλη διαδικασία της συζήτησης για το μέλλον της ε, ΟΝΕ. Στη σχετική έκθεση, η οποία είχε εκπονηθεί κατά τελευταία φορά, ε, εστιάσαμε στις μελλοντικέ εξελίξεις ε, που θα μπορούσαν να προκύψουν σε σχέση με την ΟΝΕ και σε εκείνη την έκθεση θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι θεωρήσαμε σημαντική την φάση κατά την οποία θα ξεκινήσει η διαδικασία της εκ νέου σύγκλησης, αν θέλετε. Είναι σημαντική λοιπόν ε, αυτή η φάση γιατί στο πλαίσιο τη ε, κρίση υπήρξε μια απόκληση σε ό,τι αφορά τι τοποθετήσει και τι πολιτικέ μεταξύ των κρατών μελών. Πράγμα βέβαια το οποίο κατέστησε πιο δύσκολη ε, την λήψη κοινών μέτρων σε επίπεδο Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Και βέβαια νομίζω πω αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν θέλουμε μια κοινή πολιτική θα πρέπει να υπερβαίνουμε τις διαφορές μας και να ε, προβαίνουμε σε πραγματικά κοινά μέτρα. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις τα ζητήματα είναι πιο βαθιά, δεν είναι απλά διαφορές απόψεων, υπάρχουν δηλαδή διαρθωτικού διαθροτική φύση προβλήματα και εκεί χρειάζεται να επιτύχουμε περισσότερη σύγκληση. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να εδραιώσουμε, αν θέλετε, να κατοχυρώσουμε τα όσα έχουμε. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση, η οποία δημιουργήθηκε σε συνέχεια της ε, χρηματοπιστωτικής ε, κρίσης. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τη εδραίωση αυτή τη Τραπεζική Ένωση και στο πλαίσιο ε, της Προεδρία Προεδρίας στο ΕΚΟΦΑΝ αναφέραμε το τι ακριβώ θα πρέπει να γίνει ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι μέσω τη Τραπεζική Ένωση, προκειμένου ακριβώ, να καταστεί πιο εύρωστη η Τραπεζική Ένωση και να μπορέσουμε να κατανείμουμε καλύτερα του κίνδυνου. Οι κεφαλαγορέ τώρα και εδώ μπορούμε να επιτύχουμε περαιτέρω πρόοδο. Μία σειρά από προτάσει έχουν ε, τεθεί και από την πλευρά του Κοινοβουλίου και από την πλευρά του Συμβουλίου. Ενδεχομένω θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε την όλη συζήτηση για να πετύχουμε πρόοδο και νομίζω πως θα μπορούσαμε να επιτείνουμε τη συνεργασία μας σε ό,τι αφορά το θεματολόγιο για την Ενεργειακή Ένωση και την Ψηφιακή Ένωση. Οπότε υπάρχουν μία σειρά από θεματικά ε, παιδεία στα οποία θα μπορούσαμε να επιτύχουμε περισσότερο πρόοδο και τα οποία με τη σειρά θα μας επιτρέψουν να εμβαθύνουμε περισσότερο την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Μπερές για τους σοσιαλιστές. Η ερώτησή μου είναι συνέχεια του συντονιστή, της ερώτησης του συντονιστή του ΕΛΚ στη Λευκή Βίβλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ο Ζαν Κλοντ Ιουνκέρ έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει. Δηλαδή απευθύνθηκε στα κράτη-μέλη για να μάθουμε τι ακριβώς θέλουν ε, να κάνουν από κοινού. Και ήταν σημαντικό στα πλαίσια των εθνικών εκλογών που επρόκειτο να διεξαχθούν. Οι πρώτες εκλογές έγιναν στις χώρες, στη χώρα σας δεν μπορώ λοιπόν να αντισταθώ ε, στον πειρασμό να σας θέσω την ερώτηση. Πώς αναλύεται την απάντηση που η δική σας ε, χώρα θα δώσει στην Λευκή Βίβλιο του Ζων Κλοντ Γιούνκερ με βάση και τα αποτελέσματα των εκλογών που μόλις έγιναν. Επίσης, είσαστε εκείνος που προκαλέσατε την έκθεση των πέντε προέδρων. Δεν έχουμε την ίδια βέβαια ερμηνεία του. Νομίζω στη δεύτερη φάση, πριν το 2017, Πολλά μπορούσαν ήδη να γίνουν στα πλαίσια των συνθήκων. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε, σίγουροι ότι έχουμε αξιοποιήσει πλήρω το δυναμικό το, της έκθεσης των ε, πέντε προέδρων. Χάνουμε λοιπόν χρόνο. Θα πρέπει να θέσουμε λοιπόν την ερώτηση πώς θα καλύψουμε κάπως αυτή την καθυστέρηση για να διορθώσουμε τα πράγματα. Και κατόπιν είπατε, αλλά δεν ήμουν παρούσα, αλλά αυτά διαβάζω, ότι ήσασταν υπέρ ενός ε, Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου με βάση την πείρα που είχατε στα πλαίσια της λειτουργίας της Τρόικα. Αλλά όπως ξέρετε, μαζί με τον ε, κύριο Μπέργκε, είμαι η συγκήτρια μιας έκθεσης που αναφέρεται σε ένα τέτοιο ταμείο, αλλά σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Θα πρέπει να υπάρχει αναγκαία δημοσιονομική ικανότητα. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δική σας θεώρηση, πώς εσείς το βλέπετε αυτό το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Ευχαριστώ, λέει ο κύριο Στα πλαίσια των υπαρχουσών συνθήκων μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Αυτό είναι το πρώτο σημείο και συμφωνώ απόλυτα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Μία είναι βεβαίως να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο. Το ESM θα μπορούσε, ο Μηχανισμός ε, ε, Σταθερότητας, δεν είναι αυτή η θέση του Eurogroup, είναι η προσωπική μου θέση, ότι θα ήταν κάτι τέτοιο επιθυμητό στο μέλλον. Πρώτα απ' όλα, γιατί έχει μεγάλη πείρα στην εφαρμογή προγραμμάτων. Βεβαίως, θα θέλαμε στο μέλλον να μην έχουμε τέτοια προγράμματα στα πλαίσια της ΟΝΕ, αλλά μπορεί να έχουμε. Οπότε θεωρώ ότι στο μέλλον θα ήταν ακριβώς καλό να έχουμε έναν ευρωπαϊκό θεσμό με την αναγκαία πείρα, τις αναγκαίες αρμοδιότητες και την αναγκαία δυνατότητα δράσης για να σχεδιάσει και να βοηθήσει την εφαρμογή προγραμμάτων σε χώρες προγράμματος. Ο ESM νομίζω είναι ο κατάλληλος θεσμός για να προχωρήσει το θέμα αυτό με τις δυνατότητες που ήδη έχει. Για τη δημοσιονομική ικανότητα τώρα. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. για να ορίσουμε τι στόχους ακριβώς θα θέλαμε. Υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις ακόμη γι' αυτό. Θα είναι ένας μηχανισμός επενδύσεων, θα μας δίνει έναν ε, δημοσιονομικό, ε, μια δημοσιονομική δυνατότητα για να αντιμετωπίσουμε ασυμμετρικές, ε, ασυμμετρικά σοκ. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ιδέες. Ασύμμετρα σοκ. Και επίσης υπάρχουν πολύ διαφορετικές ιδέες για το ποιος θα χρηματοδοτήσει αυτή την ικανότητα θα πρέπει να προκύψει από τον υπάρχοντα ενωσιακό προπολογισμό. Θα πρέπει να υπάρξουν νέοι πόροι και από πού. Και υπάρχουν ε, πολύ σοβαρά πολιτικά θέματα γύρω από όλα αυτά, στα οποία δεν έχουμε ακόμη απάντηση. Είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει σε μια μεταγενέστερη φάση της ανάπτυξης της ΟΝΕ. Ενώ στα πλαίσια των συνθήκων που έχουμε πρέπει να πιέσουμε για να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό ακόμη υπερβάως. Ευχαριστώ. Αν ο ESM γίνει Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, δέχεστε ότι πρέπει να γίνει στα πλαίσια των ενωσιακών θεσμών. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό θέμα. Και ε, δεν μπορώ να ε, μην ξαναρωτήσω πώς θα συμβάλλει η χώρα σας ε, στην απάντηση στα ερωτήματα που θέτει ο Ζαν Κλοντ Juncker στα πλαίσια του, της Λευκής Βίβλου. Κοιτάξτε, όσο αναπτύσσεται περαιτέρω ο μηχανισμός σταθερότητας, θα πρέπει να γίνει ένας ε, κανονικός ευρωπαϊκός θεσμός που θα λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η εξελικτική διαδικασία και αυτή είναι η λογική κατάληξή της από πλευράς αρχής. Αλλά εδώ πάλι εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Τώρα, τι μπορεί να κάνει η Ολλανδική κυβέρνηση. Ε, είναι δύσκολο θέμα για να απαντήσει ένα υπουργό ε, που απλώ ασκεί τα καθήκοντά του. Με ρωτάτε ω ε, Ολλανδό υπουργό. Όπω ξέρετε, αυτή τη στιγμή απλώ ασκώ καθήκοντα. Ορισμένοι ε, είπαν ότι είναι φιλοευρωπαϊκή έκβαση των Ολλανδικών εκλογών. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρο. Όχι τόσο σίγουρο. Αλλά δεν ξέρω τώρα πώ θα διαμορφωθεί η νέα κυβέρνηση, τι θέσει θα έχει για το μέλλον τη Ένωση. Οπότε είναι δύσκολο να προβλέψω. Πρόεδρος. Να ασχοληθούμε κυρίω όμως με τι αρμοδιότητε Προέδρου του Eurogroup. Ήταν μόνο μια παρατήρηση ως Προέδρου. επόμενο από το ECR ο κύριος Μαριά. Κύριε Ντάισεμπλουμ, ε, η Ελλάδα επί 7 χρόνια, το 2010 μέχρι σήμερα, έχει πάρει 240 δισεκατομμύρια ευρώ ως δάνεια. Θα περίμενε κανείς να έχει μια ανάπτυξη χώρα και όμως έχουμε στρατιέ φτωχών και ανέργων. Το πρόγραμμα έχει αποτύχει γιατί πολύ απλά τα δανεικά πήγαν για να πληρώσουν τα παλιά δανεικά. Ξαναπήγαν πίσω στι έπε των δανειστών. Ταυτόχρονα απαιτείται ως Eurogroup καινούρια μέτρα με μειώσεις των ε, συντάξεων, με μείωση του αφορολογήτου, που σημαίνει ακόμη μια πιο σκληρή πολιτική. Σας ρωτάω λοιπόν πολύ απλά το εξής από το τρίτο δανειακό πακέτο των 86 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 19,5 δις ευρώ, διότι 25 δις θα πήγαιναν στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, χρησιμοποιήθηκαν μόνο 4,5 δις, επομένως περισσεύουν 19,5 δις ευρώ. Οι ερωτήσεις μου είναι απλές. Πρώτον, συμφωνείτε να δοθεί ένα ποσό της τάξης των 14 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων τα οποία έχουν υποστεί ζημία λόγω του PSI. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, με τη ρευστότητα αυτή θα ενισχυθεί το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, δεν θα γίνουν οι μειώσεις στις ε, συντάξεις που απαιτείται και επενδυόμενα αυτά τα χρήματα θα δώσουν 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στο ασφαλιστικό σύστημα. Ερώτηση δεύτερη. Από το ποσό το οποίο επίσης περισσεύει των 19,5 δις ευρώ να χρησιμοποιηθούν 4,5 δις ευρώ για τη δημιουργία ενός ταμείου για τα κόκκινα δάνεια, το οποίο θα ενισχύσει αυτή τη στιγμή τους δανειολήπτες, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσει ακριβώς επειδή μειώθηκαν τα εισοδήματά τους. Και έτσι θα στηριχθεί και η δυνατότητα των τραπεζών να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό που ονομάζουμε κόκκινα δάνεια. Είναι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις αυτές και θα ήθελα συγκεκριμένες απαντήσεις στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στα ελληνικά λοιπόν, το κατάλαβα την ελληνικά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι ε, τα μέγιστα ποσά στα οποία έχουν δοθεί στα πλαίσια του τρίτου προγράμματος δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου και ελπίζω δεν θα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε όλα. Πρέπει να δούμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί είναι διαθέσιμη η πόρη αυτή. Θα πρέπει όμως να συνειδητοποιήσετε ότι όλα αυτά τα χρήματα θα περάσουν μέσω δανείων στην Ελλάδα και θα αποτελέσουν τμήμα του δημόσιου χρέους που είναι ήδη υψηλό. Κοινό λοιπόν στόχο θα πρέπει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό, χρησιμοποιώντα όσο δυνατόν λιγότερα από τα χρήματα αυτά, από τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Το πρώτο επιχείρημα που θα χρησιμοποιήσω λοιπόν είναι ότι στόχο δεν θα πρέπει να είναι να χρησιμοποιήσουμε το πλήρω των πόρων αυτών, αλλά να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα και να κάνουμε την ελληνική οικονομία να ανακάμψει χρησιμοποιώντα όσο δυνατόν λιγότερα από τα χρήματα αυτά γιατί όπω σα είπα, όσο περισσότερα χρήματα χρησιμοποιούμε, τόσο αυξάνεται το δημόσιο χρέο τη χώρα. Όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, ήδη από το Eurogroup του Φεβρουαρίου, είναι να δώσουμε λιγότερη έμφαση στη λιτότητα, λιγότερη έμφαση σε περαιτέρω περικοπές δαπανών και ανταυτού να ασχοληθούμε πραγματικά με πιο βαθιές μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να κάνουν το σταξιωτικό σύστημα πιο βιώσιμο, πιο βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Και μέρος συμφωνίας άλλωστε είναι ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί το σύστημα αυτό με ένα καλύτερο σύστημα συνταξιδοτικό το οποίο να λειτουργεί ορθώς και θα πρέπει να λειτουργεί παράλληλα. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που εξαρτώνται από το εξωτικό σύστημα ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας το οποίο να λειτουργεί σωστά, να λειτουργεί ορθά. Όσον αφορά τώρα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών έγινε ήδη στα τέλη του προηγούμενου έτους και ένα μέρος των τραπεζών ανακαιροποιήθηκαν χρησιμοποιώντας λιγότερα χρήματα από ό,τι είχαμε προβλέψει, το οποίο είναι θετικό, διότι υπήρχαν ιδιώτες επενδυτές δηλαδή, οι οποίοι ήταν τελικά σε θέση να επενδύσουν σε αυτές τις τράπεζες και ουσιαστικά γίνανε μέτοχοι στις τράπεζε αυτέ, Καταφέραμε λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο να ανακεφαλοποιήσουμε τι τράπεζε αυτέ, και κατά αυτόν τον τρόπο εν μέρη ρυθμίσαμε μέσω ιδιωτικών πόρων το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και προτιμούμε γενικά να χρησιμοποιούμε ιδιωτικού πόρου ή δυνατόν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Εφόσον λοιπόν το πακέτο των 86 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν το χρησιμοποιούμε κατά 25%, δηλαδή παίρνουμε 25% λιγότερο κεφάλαιο, για ποιο λόγο τα μέτρα που συνοδεύουν το δάνειο επιβάλλονται στο 100% και ίσως και στο 120%. Το σωστό θα είναι να μειώσετε τα μέτρα και τις απαιτήσει κατά 25% εφόσον παίρνουμε 25% λιγότερο κεφάλαιο από το δάνειο. Ευχαριστώ. No, I'm sorry, I don't follow that argument. Συγγνώμη, δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτό το επιχείρημα. Δεν συμφωνώ, δεν μου φαίνεται λογικό. Η δική σας η προσέγγιση είναι ότι έχουμε τα χρήματα αυτά, έχουμε δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουμε. Εγώ σας λέω ότι θα πρέπει να δανειστείτε όσο το δυνατόν λιγότερο, γιατί όσο περισσότερο δανειζόμαστε, τόσο αυξάνεται το δημόσιο χρέος. Αν μπορούμε λοιπόν να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα, αν μπορεί η ελληνική οικονομία να ανακάμψει, και δεν έχει συμβεί αυτό ακόμα, είμαι ο πρώτο που το παραδέχομαι. Αν καταφέρουμε να το κάνουμε χωρί να χρησιμοποιήσουμε το σύνολο των 86 δισεκατομμυρίων, αυτό θα είναι θετικό νέο για την Ελλάδα. Ναι, αλλά θα πρέπει να μειώσετε τότε κατά 25% και τα μέτρα που θέλετε να επιβάλλετε στη χώρα. Αυτό, αυτή θα είναι η λογική προσέγγιση. Πρόεδρο, καλύψτε το χρόνο που σα αναλογούσε. Α περάσουμε τώρα στου φιλελεύθερου. Νίλ Στόρετ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουν γίνει πολλές διαπραγματεύσεις μεταξύ των διαφορετικών ε, τελικά ε, φορέων ως προς το ποιος έχει δίκιο σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Ελλάδας και βέβαια ειδικότερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Επιτροπή έχουν ε, ε, αναδειχθεί ε, ιδιαίτερα σε αυτήν τη συζήτηση. Θα μπορούσατε εσείς να μας πείτε σήμερα ποιος έχει τελικά δίκιο για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Και ένα δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω. Είπατε, έχουμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία εφαρμογής. Εμένα μου ακούγεται πολύ αμφίσιμη αυτή ε, διατύπωση. Δηλαδή πότε θα ολοκληρωθεί τελικά αυτή η διαδικασία εφαρμογή. Μήπως είναι φημισμός αυτό που είπατε, ότι ουσιαστικά δεν ε, συμβαίνει τίποτα και απλώ δεν θέλετε να αναλάβετε καμία ευθύνη. Κύριε Στέσσα, αν θέλετε να αξιολογήσετε τα προγράμματα αυτά προς την Ελλάδα, θα πρέπει να επιστρέψετε λίγο ε, στην κατάσταση πριν από την κρίση και να δείτε πού ξεκίνησαν οι ανισορροπίες και ποια ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα πριν από την κρίση. Όταν δηλαδή αποκαλύφθηκαν εκείνα τα δημοσιονομικά μεγέθη, ε, είδαμε ότι από την αρχή της κρίσης είχαμε δημοσιονομικό έλλειμμα 15% ε, και το δημόσιο χρέος είχε φτάσει ήδη σχεδόν στο 100%. Οπότε τα όσα ακούγονται σήμερα, ω προς το ότι δηλαδή τα συναπτά προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα δεν λειτουργούν, θα πρέπει να ρίξει μια ματιά στο πού βρισκόταν η Ελλάδα κατά την έναρξη τη κρίση Και έχουν γίνει πολλά ε, σημαντικά βήματα στην Ελλάδα με οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Ναι, η εφαρμογή υπήρξε αργή, αλλά συνεχίζει να σημειώνεται πρόοδο και γενικά τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση, δηλαδή από ένα έλλειμμα που ξεκινήσαμε τη άξιου 15% αλλά από την άλλη πλευρά, βέβαια, η οικονομική ανάκαμψη επιβραδύνθηκε ξανά και ξανά λόγω αβεβαιότητα, πολιτική αστάθεια, έλλειψη εμπιστοσύνη και αναλήψεων ε, γενικά των, ε, των χρημάτων από τι ελληνικέ τράπεζε και ενδεχομένω τη μεταθέση στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν η όλη διαδικασία εφαρμογή των προγραμμάτων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Και βέβαια, ίσω αυτή η διαδικασία να είναι μια συνεχή διαδικασία που δεν ολοκληρώνεται ποτέ για καμία χώρα. Πρέπει δηλαδή να παρακολουθούμε και να βελτιώνουμε σύγχρονου του τρόπου με του οποίου λειτουργούμε σε επίπεδο και διοικητικό. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στην Ελλάδα και θα χρειαστούμε ακόμα πολλά χρόνια για να βελτιώσουμε, να ενισχύσουμε ε, του οικονομικού φορεί, τι σχετικέ δομέ, προκειμένου πραγματικά η Ελλάδα να έχει ανακάμψει πλήρω. Όμω θεωρώ ότι είναι εφικτό. Ναι, μπορεί να γίνει. Και έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από τη ελληνική κυβέρνηση. Δεν είμαι κοινικό εδώ σε αυτά που λέω. Έχετε ακόμα ένα λεπτό και 45 δευτερόλεπτα. Ναι, σε ό,τι αφορά ε, την διαφορά απόψεων μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Επιτροπής σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Δεν μου απαντήσατε. Φαντάζομαι πω ο διάλογο μεταξύ αυτών των δύο φορών θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Δηλαδή το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο είναι πιο απεσιόδοξο εντό εισαγωγικών από την Επιτροπή. Στα τρία πρώτα τρίμηνα είχαμε διαπιστώσει πράγματι ε, οικονομική ανάπτυξη, οπότε είχε δίκιο η Επιτροπή, αλλά στο τελευταίο ε, τρίμηνο αποδείχθηκε ότι η Επιτροπή είχε άδικο και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο είχε δίκιο, γιατί είχαμε αρνητική ανάπτυξη. Οπότε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακόμα σε μια εξαιρετικά ασταθή, αβέβαια αν θέλετε, ανάπτυξη. Οπότε εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι να δημιουργήσουμε σταθερότητα πολιτικά σε ό,τι αφορά τι διάφορε πολιτικέ που εφαρμόζουμε, προκειμένου να αρχίσει να ενισχύεται και να ανοίγει η οικονομία. Και αυτό βέβαια χρειάζεται και πολλή εμπιστοσύνη από πλευρά των επενδυτών, η οποία ακόμα δεν είναι τόσο ισχυρή. Ευχαριστώ, λέει ο πρώτο επόμενο ομιλητή, τον οποίο ευχαριστώ και ο καλύτερο για τα γενέθλιά του, της ευχές μας, ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Έχετε το λόγο για την ΚΟΥΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τις ευχές. Ελπίζω να ακούσω καλά νέα και από τον Γερούν Ντάισελμπλουμ για τη χώρα μου, την Ελλάδα. Συμφωνώ μαζί σας ότι έχει τεράστια σημασία η υλοποίηση αυτού που χθες συμφωνήσατε στο Eurogroup. Εκφράσατε όλοι, όπως δηλώσατε, μια ισχυρή πολιτική βούληση να ολοκληρωθεί γρήγορα η δεύτερη αξιολόγηση. Γιατί η παράταση αυτής τη εκκρεμότητα δημιουργεί αβεβαιότητα, βλάπτει την ελληνική οικονομία, βλάπτει κυρίως τους ασθενέστερους Έλληνες, τους άνεργους που περιμένουν μέσα από την ανάπτυξη να μειωθεί η ανεργία. Οι προβλέψεις για το 17, το 18 και το 19 και τη Κομισιόν και του IMF και του Eurogroup είναι θετικές, άρα πρέπει να επιταχύνεται αναφέρατε στην εισαγωγική σας ομιλία ότι ένα από τα μεγάλα εκρεμή θέματα και σωστά αποφασίσατε να βάλετε μπροστά τα μεγάλα και να μείνετε να δουλέψετε εδώ στις Βρυξέλλες για την επίλυσή τους μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες ή εβδομάδες. Ένα από τα μεγάλα θέματα είναι οι συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Αναφερθήκατε στην ανάγκη να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα το ευρωπαϊκό κεκτημένο, οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Σας ερωτώ, έχει υπάρξει ένα πόρισμα μιας ομάδας ειδικών την οποία την ορίσατε. Εσείς οι δανειστές τους αναθέσατε την εντολή, έχουν καταθέσει ένα πόρισμα το οποίο ζητάει την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στην Ελλάδα και των κλαδικών. Η ερώτησή μου είναι, εσείς προσωπικά που ανήκετε και στο εργατικό κόμμα, είστε σοσιαλδημοκράτης, τι θέση έχετε για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στην Ελλάδα. Ποια είναι η στάση σας απέναντι σε αυτό το πόρισμα. Και επειδή ακούω ότι το IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λέει δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, δεν καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και δεν μας ενδιαφέρει το πόρισμα των ειδικών που και οι ίδιοι συμφώνησαν. Σας ερωτώ, τι στάση θα πάρετε εσείς σε αυτό το θέμα. Καταρχάς και πάλι χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Τώρα, ως σοσιαλδημοκράτης είμαι υπέρ των συλλογικών διαπραγματεύσεων και πιστεύω ότι όντως είναι βέλτιστη η ευρωπαϊκή πρακτική. Αυτό που συμφωνήσαμε με την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2015 ήταν ότι η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας που είχε ήδη εφαρμοστεί τότε θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να μην αντιστραφεί και ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια ομάδα εμπειρογνώμων για να συμβουλεύσει την Ελλάδα για το μέλλον, την εξέλιξη της αγοράς εργασίας και των θεσμών της. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων ομόφωνα κατέληξε ότι οι συλλογικέ διαπραγματεύσει είναι νοσιακή βέλτιστη πρακτική και θα πρέπει να επανέλθει στην Ελλάδα. Τώρα ο ακριβής σχεδιασμός της ε, σχεδιασμό των διαπραγματεύσεων θα πρέπει βέβαια να εξεταστεί. Σε ορισμένε χώρε υπάρχουν κάποια κριτήρια αντιπροσωπευτικότητα για τι συλλογικέ διαπραγματεύσει. Οι διαπραγματεύσει πρέπει να γίνονται από αντιπροσωπευτικού εταίρου. Αυτά τα κριτήρια πρέπει και πιστεύω ότι θα συζητηθούν με του θεσμού. Συζητώνται αυτή τη στιγμή. Αλλά η γνώμη τη ομάδα εμπειρογνωμόνων ήταν απόλυτα σαφή για το θέμα αυτό. Ας δούμε λοιπόν ε, πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ναι, αλλά και εσείς λοιπόν είπατε θέλετε και άλλη απάντηση. Στο, στο οποίο υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους Ευρωπαίους δανειστές και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυση του χρέους. Και συμφωνήσατε να ληφθούν μετά το τέλος του προγράμματος αλλά και να προσδιοριστούν τώρα για να διευκολυνθεί η απόφαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ενώπιση της Αρινής Συνόδου. Η ερώτησή μου είναι, εσείς πιστεύετε ότι πρέπει σε αυτό το θέμα να κάνει κάποιες υποχωρήσεις το Eurogroup προς την πλευρά των απαιτήσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή μόνο για τις συλλογικές συμβάσεις συζητάτε τις αιμονές του Δουνουτού. So, I get 10 seconds for a completely new topic. Um, δευτερόλεπτα για εντελώ καινούργιο θέμα, εντελώ δύσκολο. πρόθεσμα μέτρα για το χρέο. Θα πρέπει να εφαρμοστούν ε, φυσικά μετά το τέλο του προγράμματο με δύο προποθέσει. Πρώτον, το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί επιτυχώ. Η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή να ε, εφαρμόσει τα συμπεφωνημένα. Και δεύτερον, να θα εφαρμοστεί στο βαθμό που θα χρειαστεί. Και θα κάνουμε έναν απολογισμό τη κατάσταση ε, το δεύτερο μέρο το δεύτερο εξάμεινο 18 για να δούμε ποια είναι η βιωσιμότητα. Στη συμφωνία πέρυσι το Μάιο ήδη ε, σκιαγραφίσαμε κάποια μέτρα που θα μπορούσαμε να πάρουμε. Ίσως το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ να επανέλθει και να πει ότι δεν είναι επαρκώς συγκεκριμένα τα μέτρα αυτά, πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν περισσότερο, εντάξει, να το συζητήσουμε, να δούμε τι περαιτέρω διευκρινήσεις μπορεί να χρειαστούν, αλλά σε τελευταία ανάλυση τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν μετά τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή στα μέσα του 18, το δεύτερο εξάμεινο με βάση την μελέτη ε, βιωσιμότητας του χρέους που θα γίνει τότε. Την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους. Βεβαίως, αν χρειαστεί, δεσμευόμεθα να κάνουμε συζήτηση τις επόμενες εβδομάδες και μήνες με το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ. Αλλά τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν το δεύτερο μισό του 18. Αυτό δεν αλλάζει. Ορίστε, πήρατε ένα λεπτό παραπάνω λόγω των γενεθλίων σας. Ερνέσουρ Ουρτασούν. Σας ευχαριστώ κύριε Ντάισεπλουμ. Τρία πράγματα. Πρώτον, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Παπαδημούλης πριν από λίγο, Μπορούμε λοιπόν βεβαίωσουμε ότι υπάρχει δέσμευση από τη δική σας την πλευρά ως πρόεδρου του Eurogroup ότι όντως τάσεστε υπέρ της επανένταξης των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα και ότι θα λαφθεί υπόψη το πόρισμα της ομάδας εμπειρογνωμόνων είναι πολύ σημαντικό να φανεί ότι δεσμεύεστε εσεί γι' αυτό απέναντι στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Θα ήθελα από αυτού μία απάντηση από εσά. Δεύτερον, στα πλαίσια του Eurogroup μιλήσατε για τη βιωσιμότητα των στεξιδοτικών ταμείων. Αν πάμε στην Ελλάδα, τα τελευταία, το τελευταίο χρόνο οι μεταρρυθμίσεις οδήγησαν σε μια κατάσταση όπου ενώ στο παρελθόν χρειαζόμασταν τέσσερις, ταξιούχους, τέσσερις εργαζόμενους για ένα συνταξιούχο, τώρα χρειαζόμαστε δέκα εργαζόμενους για να υποστηρίξουν τη σύνταξη ενός συνταξιούχου. Νομίζω λοιπόν ότι και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ιδίως όταν μας λέτε ότι θα χρησιμοποιήσετε benchmarking για τις συντάξει πλέον στην Ευρώπη. Και τρίτον, σε μία δήλωση που κάνατε πρόσφατα στην Frankfurter Allgemeine Zeitung. Είπατε είπατε κάτι που δημιούργησε σκάνδαλο σε καποια κρατημέλη όταν είπατε, αναφερόμενο στην κρίση δηλαδή, ότι δεν μπορούμε να καταναλώνουμε χρήματα σε αλκοόλ και σε γυναίκες και μετά να ζητάμε χρήματα δανεικά. Και το είπατε αυτό αναφερόμενος φαντάζομαι σε βόρειες χώρες και σε νότιες χώρες κάνοντας μια αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο. Τι ακριβώς έχετε να μας πείτε ως προς αυτό και σε σχέση με την επανυποψηφιότητά σας για το Eurogroup. Όσον αφορά τις λογικές διαπραγματεύσεις, τα πράγματα είναι σαφή, το ξέρει αυτό και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θέλουμε μια πλήρη συμφωνία πολιτικής, μια δέσμη μέτρων η οποία θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ θεσμών και Ελλάδας, ένα πλήρες πλαίσιο συμφωνίας όπου θα περιλαμβάνει και μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή συμφωνία αυτή προκειμένου να υπάρχει εμπιστοσύνη και στο Eurogroup και στα πλαίσια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και μέρος συμφωνίας θα πρέπει να είναι και συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η προσωπική μου τοποθέτηση και άποψη. Δεύτερον, όσον αφορά την βιωσιμότητα των στεξωτικών συστημάτων. Το στεξωτικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο. Αν βελτιωθεί όμω η οικονομία και αυξηθεί ο ρυθμό των εργαζομένων, τότε αυτό προφανώ βοηθά τη βιωσιμότητα των στεξωτικών συστημάτων. Αλλά μακροπρόθεσμα βλέπουμε ότι το στεξωτικό σύστημα βαρύνει πολύ τα δημόσια οικονομικά και τα βαρύνει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή ακόμα. Επομένω, δεν μπορούμε να πούμε ότι επί του παρόντο έχουμε μια βιώσιμη κατάσταση όσον αφορά τα αξιωτικά συστήματα, ούτε από οικονομική πλευρά, ούτε από πλευρά δημοσιονομική, δηλαδή βιωσιμότητα δημόσιων δαπανών. Τρίτον, η παρατήρηση που έκανα, την αποσαφηνίσω, τι σημαίνει για μένα αλληλεγγύη. Είμαι σοσιαλδημοκράτη, Εκτιμώ πάρα πολύ την αρχή τη αλληλεγγύη, λοιπόν. Στα πλαίσια μια κοινωνία και στα πλαίσια τη Ευρώπη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη σημαίνει και δεσμεύσει, υποχρεώσει και καταβολή προσπαθειών προκειμένου να κάνουμε κάθε τι το δυνατό σε ατομικό και εθνικό επίπεδο προκειμένου να ενισχύσουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Και αυτό επίση και σε κοινωνικού και οικονομικού όρου. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ανάληψη ευθυνών προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, επί το οποίο συμφωνήσαμε πρόσφατα. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση τη εθνική οικονομία, δηλαδή να γίνουν οι απαραίτητε μεταρρυθμίσει, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι απαραίτητε διορθώσει και προσαρμογέ στην οικονομία, προκειμένου κάθε χώρα να είναι ισχυρή και εύρωστη. Εφόσον λοιπόν γίνουν όλα αυτά και εφόσον αληφθούν όλε αυτέ οι ευθύνε, πιστεύω ότι ε, η αρχή της αλληλεγγύης προφανώς θα πρέπει να υφίσταται και η ελεγγύη θα πρέπει να είναι διαθέσιμη. Αυτό είναι το σχόλιο που έκανε και στην περίφημη αυτή συνέντευξη και αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Ζητάτε όμως ε, συγγνώμη για όλα αυτά τα οποία είπατε, ότι οι νότιε χώρες έχουν καταναλώσει χρήματα σε αλκοόλ και σε γυναίκες. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Θέλετε να σας διαβάσουμε πώς τη δήλωσή σας πραγματικά μου κάνει εντύπωση ότι για κάποιο λόγο διέρευσε κατά αυτόν τον τρόπο στον ισπανικό τύπο. Αυτό το οποίο είπα σαφώ είναι ότι η ελεγγύη θα πρέπει να συνοδεύεται με ευθύνε και ανάληψη υποχρεώσεων και ευθυνών. Διαφορετικά η ελεγγύη αυτή δεν θα είναι βιώσιμη. Δεν μπορούμε να έχουμε υποστήριξη για την αρχή τη ελεγγύη αν παράλληλα δεν έχουμε καταβολή προσπαθειών και ανάληψη ευθυνών από όλε τι πλευρέ. Έχω δέκα δευτερόλεπτα, διαβάζω τη δήλωσή σας. Δεν μπορεί κανείς να καταναλώνει όλα τα χρήματά του σε ποτά και σε γυναίκες και μετά να ζητά χρήματα και δανεικά. Ζητάτε συγγνώμη για κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Και ε, μη μου διαβάζετε εσείς τη δήλωσή μου, γιατί εγώ τη γνωρίζω καλύτερα από εσά. Εγώ έκανα τη δήλωση αυτή, γνωρίζω ακριβώς τι είπα. Εσείς πρέπει να καταλάβετε λοιπόν ότι αν θέλετε να υπάρχει μια πολιτική υποστήριξη και αλληλεγγύη παντού στην Ευρωζώνη και σε οποιαδήποτε κοινωνία, τότε παράλληλα θα πρέπει να γίνεται και μια συζήτηση για τις δεσμεύσεις που πρέπει όλοι να αναλάβουν και τις ευθύνες που πρέπει όλοι να αναλάβουν, προκειμένου από την άλλη πλευρά να έχετε και την ελληνική των υπόλοιπων εταίρων. Αναλώστε το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας. Ο κύριος Άνεμανς έχει το λόγο, παρακαλώ. Ik weet wel dat het voorzitterschap van de Eurogroep eh, niet echt iets is dat democratisch verloopt. Ο oh, eh, πρόεδρος ε, ε, του Eurogroup ε, δεν εκλέγεται βέβαια με ιδιαίτερα δημοκρατικό τρόπο, πράγμα βέβαια το οποίο δεν συζητείται συχνά εδώ στο Κοινοβουλίο, αλλά θα ήθελα να αναφέρω ότι αναφέρθηκε στον αδικό τύπο ότι ε, το Eurogroup αποφάσισε να συνεχιστεί η θητεία σας κανονικά ως ε, πρόεδρος ε, του Eurogroup ενώσο είσαστε υπουργό Οικονομικών των κατοχωρών. Οπότε αποτελεί προϋπόθεση τυπική το να είναι κανείς υπουργό Οικονομικών για να παραμείνει πρόεδρος του Eurogroup. θα συνεχιστεί δηλαδή η θητεία σας και δικαιούστε να συνεχίσετε τη θητεία σας ή όχι. Ένα δεύτερο ερώτημα. Εδώ στον τύπο αναφερόταν ότι υπάρχει ένα επιχείρημα υπέρ του να παραμείνετε σε αυτή τη θέση του Προέδρου και ότι θα χρειαστεί να προβείτε και σε δύσκολε διαπραγματεύσει μέσα στου επόμενου μήνε σε ό,τι αφορά το τρίτο πρόγραμμα για την Ελλάδα. Εσείς, όταν διαπιστώνετε ως σοσιαλδημοκράτης πως η πολιτική λιτότητα στην οποία εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη ουσιαστικά έχει αντίκτυπο σε διάφορες χώρες και στο πολιτικό για παράδειγμα επίπεδο, το οποίο συνέβη και στη δική σας χώρα αλλά και για παράδειγμα στην Ελλάδα, δεν ε, δικαιολογεί το να επιθυμείτε κι εσείς από την πλευρά σας να ε, μην συνεχίσετε ως πρόεδρος του Eurogroup και να δώσετε τη δυνατότητα σε κάποιον άλλο να αναλάβει ως πρόεδρος ώστε να βοηθήσει στην επίλυση των ε, προβλημάτων της Ελλάδας. Μίσος δηλαδή δεν φάνηκε και αυτό στις ε, εκλογές της δικής σας χώρα. Ναι. Και κοιτάξτε, η θητεία μου συνεχίζεται κανονικά. Ακόμα ε, δεν έχει σχηματιστεί νέα κυβέρνηση στι κατοχώρε, οπότε δεν έχει τεθεί ακόμα προ το αν θα συνεχίσω ή όχι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μέλλον και τι θα συμβεί από εκεί και μετά, αυτό εξαρτάται από τους υπουργούς του ε, υπουργού του Eurogroup. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα για την Ελλάδα, ίσως ε, το δικό σας συμπέρασμα ε, είναι ότι το αποτέλεσμα των ε, εκλογών στις κάτω χώρες είναι ότι ουσιαστικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε εντελώ διαφορετικό τρόπο το ζήτημα της δημοσιονομικής πειθαρχίας σας επιμέλειας, αλλά η δική μου εντύπωση είναι διαφορετική. Ότι δηλαδή ουσιαστικά το συμπέρασμα είναι ότι ακριβώς θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί στο μέλλον σε ό,τι αφορά τέτοιου είδους ζητήματα δημοσιονομικής επιμέλειας. Πρόεδρε, δεν ε, είπα ακριβώς αυτό. Εγώ είπα ότι δεν έχει νόημα για τους ε, σοσιαλδημοκράτες ε, το να εφαρμόζουν τέτοιου είδους πολιτικές, να προσυπογράφουν τέτοιου είδους πολιτικές. Είναι μια περίοδος νίκη και σας λέω ότι αυτό δηλαδή έχει αντίκτυπο και στο πολιτικό επίπεδο και στην Ελλάδα. Μήπως λοιπόν δεν έχει νόημα να συνεχίσετε να έχετε αρμοδιότητες για τέτοια ζητήματα. Σε ό,τι αφορά ε, την ανάλυση σε ό,τι αφορά ε, που κάνατε σε σχέση με το αποτέλεσμα των ανδικών ε, εκλογών. Δεν έχετε δίκιο γιατί οι σοσιαλιστές προφανώς έχασαν πολύ έδαφος. Από εκεί και μετά σας ξαναλέω οι αρμόδιοι για τον, τη λήψη της απόφασης του κατά πόσο είναι ενδεδειγμένος ένας πρόεδρος του Eurogroup ή όχι είναι υπουργοί του Eurogroup. Πρόεδρος, δεν νομίζω πως έχει νόημα το να συζητάμε εδώ θητεία του κυρίου Ντάσιμπλου, πρόεδρου του Eurogroup. Και η συζήτηση των ε, Ολλανδικών εκλογών δεν νομίζω πω θα πρέπει να γίνει εδώ. Θα πρέπει να την διεξάγετε αλλού αυτή τη συζήτηση για την LP ε, του David Coburn. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ντάισμπλουμ, είμαι σίγουρο ότι έχετε στενή σχέση εργασία με τον κύριο Μάριο Ντράγκη τη ΕΚΤΑΦ. Θα πρέπει να συνομιλείτε συχνά μαζί του Οπότε σας παρακαλώ μπορείτε να του εξηγήσετε τη σημασία του να απαντάει στις ερωτήσεις των βουλευτών. Εγώ και άλλοι συνάδελφοι από άλλες πολιτικές ομάδες του έχουμε υποβάλει μια σειρά ερωτήσεων για την ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του ρόλου του ως Προέδρου της ΕΚΤ και των προηγουμένων πράξεων του ή παραλήψεων ως κυβερνήτου της ε, διοικητού της ε, ε, κεντρική τράπεζα Ιταλία. Του το έχουμε ζητήσει ω Επιτροπή, γραπτό, προφορικά. Έχουν περάσει μήνε, Από πέρυσι δεν έχουμε ακόμη απάντηση. Εάν καταρρεύσει το Ιταλικό τραπεζικό σύστημα, τότε θα υποθούν πολλά για το ρόλο του ω διοικητού τη Κεντρική Τράπεζα. Και αυτό θα υπονομεύσει όχι μόνο το Ιταλικό τραπεζικό σύστημα, αλλά και το Ευρωπαϊκό. Και τον τρόπο με τον οποίο οι Εθνικέ Κεντρικέ Τράπεζε ε, συνεννοούνται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το να αποφεύγει να δώσει απαντήσει ε, δημιουργεί θεωρίε συνωμοσία βέβαια. Άρα προ το συμφέρον τη ε, δημοσιονομική σταθερότητα τη Ευρωζώνη μπορείτε παρακαλώ να υπενθυμίσετε στον πρόεδρο Ντράγκη όχι μόνο τι ερωτήσει που του θέσαμε αλλά και τη σημασία του να μα δώσει σωστέ απαντήσει. Και είναι ανησυχητικό αυτό γιατί οι πρόσφατες αλλαγές ε, στην διαδικασία, στους διαδικαστικούς κανόνες, θα ε, επιτρέψει ακόμη περισσότερο διαφανείς διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα συζητάνε σε κλειστέ αίθουσε που δεν θα καπνίζουν πια, θα καπνίζουν ηλεκτρονικά τσιγάρα, αλλά αυτό δεν αλλάζει την ουσία τη υπόθεση. Ο κύριο Ντάζιμπλουμ. Δεν έχω υπόψη μου αυτέ τι ερωτήσει και είμαι σίγουρο ότι δεν χρειάζεται να στείλω εγώ μηνύματα στον Ντράγκη. Νομίζω ότι το κοινοβούλιο είναι σε θέση να του αποστείλει ερωτήσει. Ναι, λέει ο κύριο Κόμπερντ, το έχουμε θέσει επανειλημμένα αυτέ τι ερωτήσει και δεν έχει απαντήσει. Γι' αυτό σα ζητάω εσά να παρέμβετε. Είναι πολύ ανησυχητικό. Θέλουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Τι είναι έχει να καθόμαστε εδώ μέσα και να θέτουμε ερωτήσει ω κοινοβουλευτικοί και να μην λαμβάνουμε απαντήσει. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με του νέου κανόνε κινείται προς ε, διοίκηση παρασκηνίων και όχι μέσω κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Εμεί φεύγουμε τώρα. Αλλά δεν θέλουμε να σας αφήσουμε και να έχουμε εδώ δίπλα στην πόρτα μας ε, μια κατάσταση ε, λυπηρή. Δεν θέλουμε η Ευρώπη να γίνει μη δημοκρατική περιοχή. Μήπως μπορείτε να κάνετε κάτι. Πρόεδρος, έχουμε σαφείς κανόνες, David, για το τι ερωτήματα θέτουμε στον πρόεδρο της ΕΚΤ Είναι σαφές είναι κανόνες που έχουν εγκριθεί από τον πρόεδρο, πρέπει να γίνει αυτή η ερώτηση και πρέπει να εγκριθεί από το Προεδρείο. Μόνο έτσι μπορούμε να θέσουμε ερωτήσει στον Πρόεδρο της ΕΚΤΑΦ και αν χρόνο λαμβάνουμε τις απαντήσεις. Και τακτικά έρχεται εδώ. Και ο Πρόεδρο ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συστημικών Κινδύνων, Συστημικών Κινδύνων και μπορούμε να του θέτουμε ερωτήματα. Ναι, αλλά δεν απαντάει ο κ. Κόμπερν. Όχι, όχι, έχουμε του κανόνε για να διαφυλάτουμε τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων. Ωραία, ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Επ' αυτού προς Σας παρακαλώ να κλείσετε το μικροφωνό σας τώρα. Για να μπορεί να ξέρει η κάμερα σε ποιον να πάει. Και τώρα θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Γιατί εγώ είμαι ο επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δάσιμπλουμ για τα όσα μας αναφέρεται σήμερα εδώ και θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα το οποίο έχει βρεθεί στο φως της δημοσιότητας επανειλημμένα και το οποίο συζητήθηκε και χθε ε, στο Eurogroup, δηλαδή τα σχέδια προπολογισμού των κρατών μελών ειδικότερα εν ώψη των υποχρεώσεων που υποκάζουν από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ε, για πρώτη φορά διαπιστώνουμε Ε, ότι υπάρχει ανάπτυξη, θετική δηλαδή, θετικός ρυθμό ανάπτυξης σε όλα τα κράτη-μέλη και αν ερμηνεύω σωστά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ε, τότε κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουν να επιτεχάνονται κάποια πλεονάσματα τα οποία ε, θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον δύσκολες περιόδους. Η Επιτροπή λοιπόν στη δική της γνωμοδότηση σε ό,τι αφορά τα σχέδια προπολογισμού των κρατών μελών διαπιστώνει ότι μόνο πέντε κράτη-μέλη συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας σταθερότητας και ανάπτυξης. Με βάση λοιπόν αυτές τις γενικές προϋποθέσεις που μόλις τώρα ανέφερα, δεν έχει φτάσει πλέον ο χρόνος να φροντίσουμε για την σωστή εφαρμογή αυτών των υποχρεώσεων από την πλευρά όλων των κρατών μελών. Και σε αυτό το πλαίσιο δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το σύνολο ε, της ε, οικονομικής κατάστασης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν θα πρέπει να δούμε πώς εφαρμόζονται τελικά οι πώ λειτουργούν οι κανόνε αυτού του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη, πώ ενδεχομένω δηλαδή είναι δυνατό ο συμψηφισμό μεταξύ πλεονασμάτων σε κάποιε χώρε με τα ελλείμματα σε άλλε. Ναι. Όντω, έχετε δίκιο ότι πέντε χώρε συμμορφώνονται πλήρω. Νομίζω ότι 7 εν γέννη συμμορφώνονται και άλλες 7 ή 6 χώρες διατρέχουν το κίνδυνο της μη συμμόρφωσης. Από τις χώρες λοιπόν αυτές ε, του ζητήθηκε να ετοιμάσουν, ε, να παρουσιάσουν και να εφαρμόσουν επιπλέον επιπρόσθετα μέτρα. Η κατάσταση βέβαια αυτή διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ορισμένες χώρες βρίσκονται στην ε, διαδικασία προετοιμασία εκπόνηση επιπλέον μέτρων. Άλλε χώρε είναι σε θέση να τα συζητήσουν ήδη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλε φορέ διαφέρει η μεθοδολογία, άλλε φορέ διαφέρουν τα δεδομένα επομένω βρίσκονται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλε χώρε έχουν ζητήσει ευελιξία. Όσον αφορά δηλαδή τι επενδύσει ή όσον αφορά τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Ευελιξία δηλαδή σε αυτού του τομεί. Είπαμε λοιπόν στο Eurogroup ότι το Μάιο βάσει των αρινών προβλέψεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό, ζητώντα από τι χώρε εκείνε που διατρέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωση να εφαρμόσουν επιπλέον μέτρα. Ορισμένε χώρε είπαν ήδη ότι θα το κάνουν αυτό. Δεν νομίζω πάντως ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να υπολογίζουμε τώρα το έλλειμμα ή το πλεόνασμα που έχουν ορισμένες χώρες και να πούμε ότι αυτό εξορροπείται και ότι αντισταθμίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Κοιτάμε πάντα το σύνολο της Ευρωζώνης και βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλήσεις ακόμα και κάθε κράτος μέλος μεμονωμένα θα πρέπει να πετύχει το μεσοπρόθεσμο στόχο του, με μεσοπρόθεσμα βέβαια. Τον Ιούνιο θα συζητήσουμε στα πλαίσια του Eurogroup, ή θέλω τουλάχιστον να συζητήσουμε, το ζήτημα του δημοσίου χρέους. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές αβεβαιότητες στην παγκόσμια οικονομία όσον αφορά την Ευρώπη. Επομένως, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτή η ανάκαμψη, ότι αυτή η οικονομική ανάπτυξη που έχουμε δει του τελευταίου μήνε θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα απόθεμα προστασία, την ικανότητα δημοσιονομική προστασία στα πλαίσια τη δημοσιονομική μα κατάσταση για να αντιμετωπίσουμε μελλοντικά προβλήματα τα οποία μα περιμένουν κάποια στιγμή στο μέλλον. Είναι σημαντικό λοιπόν οι χώρε να αρχίσουν σιγά σιγά να μειώνουν το δημόσιο χρέο του, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα βρεθούμε αντιμέτωποι με δυσκολίε να έχουμε ένα δημοσιονομικό απόθεμα το οποίο θα προστατεύσει του προπολογιού μα. Η νομισματική πολιτική έχει χρησιμοποιηθεί στο έπακρο και ελπίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί λιγότερο στο μέλλον, προκειμένου να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε το απαραίτητο δημοσιονομικό αυτό απόθεμα που θα μα προστατέψει σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε δυσκολίε στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή όμω έχουμε χρησιμοποιήσει κάθε ευελιξία στο μέγιστο. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η εξομάλυνση τη νομισματική αυτή πολιτική θα συνδυαστεί με μείωση του δημόσιου χρέου. Οι δύο αυτοί παράγοντε είναι πάρα πολύ σημαντικοί προκειμένου να καταφέρουμε να απορροφήσουμε μελλοντικού δημοσιονομικού κλειδονισμού. Σα ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ο επόμενος από τους σοσιαλιστές είναι ο Ούντο Μπούλμαν. Uh, πίστευα ότι ήταν η σειρά μου, ήταν ένα δώρο. Αλλά ε, θα προτιμούσα να μιλήσω τη γλώσσα μου. Κύριε Πρόεδρε του Eurogroup, δεν επιμένω στο θέμα της Ελλάδας γιατί θέλω να δημιουργήσω δυσχέρεια σε κανένα ή στους Έλληνες συναδέλφους, αλλά γιατί έχω την εντύπωση ότι μετά από 7 χρόνια οι 8 χρόνια που ασχολούμεθα με τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας δεν έχουμε βρει τη σωστή λύση. Και έχει γίνει θέμα της αξιοπιστίας όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά συνολικά της Ευρωζώνης και συνολικά της Ένωσης. Και ιδιαίτερα οι γείτονέ μας. Ιδιαίτερα οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις και μπλοκ με τους οποίους βέβαια και συνεργαζόμεθα αλλά και είμαστε σε ανταγωνισμό, θεωρούν ότι αυτό είναι δείγμα της πολιτικής μας αδυναμίας. Ένα πρόβλημα που αρχικά τουλάχιστον φαινόταν επιλύσιμο, ε, δεν καταφέρνουμε τελικά να το επιλύσουμε. Λοιπόν, από τις αρχές του 2017 διαπιστώνω ότι έγιναν αναλήψεις 4 δις από τις ελληνικές τράπεζες. Εσείς κύριε Πρόεδρε, Είπατε ότι υπάρχει αβεβαιότητα, ότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης, ε, πολιτικής εμπιστοσύνης, δεν υπάρχει αναγκαία προσπάθεια, αναγκαία δέσμευση. Βεβαίω πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά. Αλλά στην τελική σας ε, αποτίμηση δεν θεωρείτε ότι ακριβώς το έλλειμμα εμπιστοσύνης το οποίο οδήγησε σε αυτές τις αναλήψει σε τελευταία ανάλυση είναι αποκλειστικά ευθύνη τη ελληνική κυβέρνηση. και της ανεβλητικότητας ε, των δανειστών, οι οποίοι χάνουν τη μία από την άλλη προθεσμία, όπου κάθε φορά μας λένε θα ολοκληρώσουμε και κάθε φορά μας απογοητεύουν. Έχουμε την εντύπωση ότι το θέμα δεν είναι τα οικονομικά στοιχεία, αλλά η διάθεση των Υπουργών Οικονομικών που αποφασίζουν για τα νέα καθήκοντα, και με τι τρόπο τελικά καταλήγει αυτή η διαδικασία δεν ξέρω. Τώρα, αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα των εμπειρογνώμων τη αγορά-εργασία. Κανεί δεν ενδιαφέρθηκε για τα πορίσματά μα, μα είπαν, ούτε η Κομισιόν, ούτε το Eurogroup. Δεν θέλησαν να τα συζητήσουν σοβαρά μαζί μα. Εμεί θα θέλαμε να παίξουν ρόλο στην διαμόρφωση των ε, διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει φυσικά και οι Έλληνε να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν πλεονάσματα. Αλλά σε τελευταία ανάλυση είναι η κυρίαρχη απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Πώς θα χρησιμοποιήσει αυτά τα πλεονάσματα οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, είναι θέμα δικής τους απόφασης και δεν είναι προτεκτορά του η Ελλάδα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Ντάζιμπλουμ. Νομίζω ότι βασικά το ερώτημα που θέτεται είναι γιατί καθυστερούν τόσο πολύ τα πράγματα. Και αυτό βεβαίως θίγει την εμπιστοσύνη. Αναφερθήκατε στις ε, αναλήψει. Αν αυτό είναι ευθύνη του Eurogroup και των μελών τη Ευρωζώνης, βεβαίως και είναι. Και γι' αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα το πόσο χρονοτριβεί αυτή η αξιολόγηση. Και η ανάπτυξη που είδαμε στα πρώτα τρία τρίμηνα του έτους εξαφανίστηκε μετά και κάποιε καταθέσει που έγιναν στι τράπεζε τώρα μετατράπηκαν σε αναλήψεις. Και αυτό είναι η ανησυχία μου. Γι' αυτό προσπαθώ να βοηθήσω και το Φεβρουάριο και τι τελευταίε δύο μέρε για να υπάρξει επιτάχυνση τη διαδικασία. Ούτω ώστε να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουμε ποια είναι τα βασικά θέματα, πού έχουμε κολλήσει, Πώ μπορούμε να ξεπεράσουμε τα διέξοδα. Και ω επίπτωση όλων αυτών, τώρα οι θεσμοί και η ελληνική κυβέρνηση θα συναντηθούν εδώ στις Βρυξέλλες για να ξεπεράσουν τα διέξοδα για αυτά τα βασικά θέματα. Ούτως ώστε οι θεσμοί κατόπιν να πάνε πίσω στην Αθήνα και να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση, να την κλείσουν. Γιατί η ταχύτητα είναι θέμα ζωτικής σημασίας. Ας το κάνουμε λοιπόν αυτό επιτέλους. Τώρα, πώς αξιοποιήσαμε ε, τα πορίσματα των υπερογνωμόνων για τη μεταρρύθμιση αγοράς εργασίας, όλες αυτές οι συζητήσεις γίνονται μεταξύ των θεσμών και τη ελληνική κυβέρνηση. Το Eurogroup δεν συμμετέχει στο τραπέζι να συζητάει τη μεταρρύθμιση τη αγορά εργασία, αλλά για να σα καθησυχάσω, εγώ προσωπικά έχω συζητήσει με το Διεθνή Οργανισμό Εργασία, ο οποίο είχε συμμετάσχει με του περισσότερου εμπειρογνώμονε σε αυτή την ομάδα και με, με ενημέρωσαν για τι προτάσει του και για τον τρόπο προώθησή του. Ναι, λοιπόν, βεβαίω, του έχω μιλήσει. Παίρνω πολύ σοβαρά τα πορίσματά του, αλλά, όπω και προηγουμένω είπα, Όλα αυτά πρέπει να είναι εντό του συνολικού πακέτου πολιτική που θα συμφωνηθεί μεταξύ τη Ελλάδα και των θεσμών. Και ελπίζω να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα αυτή η συζήτηση και να υποβληθεί κατόπιν στο Eurogroup. Ευχαριστώ. Γαμπριέλ Μάτο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση για τις πολιτικές προκλήσεις και την κοινή γραμμή, αλλά μετά τη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε χθε σε μια γερμανική εφημερίδα, και την απάντηση που δώσατε σε έναν συνάδελφο, δεν μπορώ να αποφύγω να σας πω ότι χάσατε μια μεγάλη ευκαιρία, μια νέα ευκαιρία. Ήταν πολύ εύκολο για σας να ζητήσετε συγγνώμη τώρα για μια δήλωση που είναι απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Και όχι μόνο δεν το κάνατε, αλλά στα πλαίσια της αλληλεγγύης όπως το θέσατε, αυτό που κάνατε ήταν να εμένετε σε μια χιδεότητα, ε, μια επιθετικότητα, μια διάθεση να μας προσβάλλετε. Και το θέμα δεν είναι ότι το αναφέρει ο γερμανικό τύπο, ο ισπανικό τύπο. Τι είπατε εσεί σε μια γερμανική εφημερίδα. Τι μα λέτε, ψεύδετε η Frankfurter Allgemeine. Αν δεν μα πείτε αυτό, τότε ψεύδεστε εσεί. Και επιπλέον, το βασικό είναι ότι χάσατε λοιπόν μια ευκαιρία. Χάσατε μια ευκαιρία να αποδείξετε την αναγκαία ουδετερότητα που πρέπει να έχει ο πρόεδρο του Eurogroup. Αυτό το οφείλεται σε όλο το Eurogroup. Οπότε η μόνη μου ερώτηση αυτή τη στιγμή είναι εάν θεωρείτε ότι μπορείτε να συνεχίσετε να εκπροσωπείτε όλα τα κράτη-μέλη του, Euro, του Eurogroup ως πρόεδρος του. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, πολύ ενδιαφέρον ξαφνικά όταν γίνεται λόγος για αλληλεγγύη. Αυτόματα υπάρχει μια σύγκρουση και την παράθεση μεταξύ διαφορετικών περιοχών της Ευρώπης και της Ευρωζώνης. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Είπα ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζουμε τα πλαίσια, τους κανόνες με σοβαρότητα, το οποίο πρέπει να το κάνουμε βέβαια όλοι μας. Και όλη η ιδέα ότι το Eurogroup είναι χωρισμένο μεταξύ Βορρά και Νότου είναι ένα τεράστιο σφάλμα δεν συζητάμε κατά αυτόν τον τρόπο, δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο στο Eurogroup. Και όταν λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι συμφωνίε και οι κανόνε μα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, αυτό έχει να κάνει με όλου του υπουργού. Μιλήσαμε για τα σχέδια προπολογισμού, μιλούσαμε για τι χώρε εκείνε οι οποίε ενδεχομένω να παρεκκλίνουν ή κινδυνεύουν να παρεκκλίνουν. Αν δείτε τι χώρε αυτέ, δεν είναι μόνο χώρε του Νότου. Είναι χώρε που βρίσκονται παντού στην Ευρωζώνη. Επομένω, όλη αυτή η προσέγγιση του ότι ξαφνικά εγώ αναφέρομαι σε συγκεκριμένου κανόνες και συμφωνίες και λέω ότι θα πρέπει να είμαι σοβαρός, ότι πρέπει να είμαι σοβαρή απέντηση σε αυτά, ότι αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε επίθεση κατά του Νότου, αυτό είναι τεράστιο σφάλμα. Ναι, να επανέλθω. Εγώ δεν είπα ότι επιτίθεστε στον Νότο. Είπα κάτι σαφέστατο. Όταν μιλάμε για αλληλεγγύη, δεν υπάρχει καμία σύγκρουση. Αλλά δεν μιλήσατε για αλληλεγγύη. Είπατε ότι ορισμένοι είναι μεν σωστοί ή ενώ άλλοι δαπανούν τα χρήματα αυτά σε γυναίκες και ποτά. Αυτό δεν είναι αλήγη. Αυτά είναι χιδεότητες. Αυτά είναι ανέδεια. Αυτό είναι καθαρή φαλοκρατική στάση. Είναι απαράδεκτο. Και είναι απαράδεκτο να προκύπτει από τον πρόεδρο του Eurogroup. Γιατί όταν λέτε ότι εμείς στο Eurogroup στο Eurogroup συζητάτε πολλά θέματα και πολύ καλά θέματα. Αλλά ο πρόεδρος του Eurogroup σήμερα έχασε απολύτω, όχι όλη την αξιοπιστία. Ορισμένοι πίστευαν ότι είχε μεγάλη και άλλη μικρή αξιοπιστία, αλλά αυτό που έχασε οπωσδήποτε πλήρω και απόλυτα είναι η ουδετερότητα. Και αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχω διαφορετική άποψη από εσά ε, ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Γιατί ω πρόεδρο του Eurogroup γνωρίζω πολύ καλά, όπω και εσεί γνωρίζετε, ότι ο μόνος ε, τρόπος για να προχωρήσουμε ε, ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να βασιστούμε στα όσα έχουμε συμφωνήσει ε, στο παρελθόν. Όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο του μηχανισμού σταθερότητας. Να συνεχίσουμε λοιπόν με βάση αυτά που έχουμε συμφωνήσει και να είμαστε αλληλέγγυοι στο μέλλον. Να, και προκειμένου να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς αυτούς θα πρέπει να συνεχίσουμε και να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στα όσα έχουμε συμφωνήσει. Και αυτή η υποχρέωση, αυτή η δέσμευση ισχύει για όλους μας, όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτό το λέω σε όλους τους υπουργούς. Όταν συζητούμε για παράδειγμα το που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική κατάσταση, όταν ασχολούμαστε με τις δημοσιονομικές ανισορροπίες στις εκάστοτε χώρες, αναφέρομαι και απευθύνομαι σε όλα τα κράτη-μέλη. Λέω ότι θα πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τα όσα συμφωνήσαμε. Σε διαφορετική περίπτωση γινόμαστε πιο αδύναμοι από πολιτική άποψη. Ο μόνο τρόπο για να ενισχυθούμε πολιτικά είναι ακριβώ να αναλαμβάνουμε την ευθύνη και να ε, εμένουμε στα όσα έχουμε συμφωνήσει. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται για μία συγκεκριμένη χώρα, δεν πρόκειται για μία ε, ομάδα από χώρε. Και οι κάτω χώρε, για παράδειγμα, δεν κατάφεραν να συμμορφωθούν με τι υποχρεώσει του και κατά συνέπεια χρειάστηκε να, κάνουν, να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειε. Τα ίδια λοιπόν ισχύουν και για του υπολείπου. Χάσατε και τρίτη ευκαιρία. Χάσατε και τρίτη ευκαιρία, ζητήστε συγγνώμη. Και τώρα ο Πολ Τάγκ. Πολ! Α, είχε φύγει. Α, μου λείψες, γιατί δεν σε είδα στη θέση σου. Θα μιλήσω στα Ολλανδικά, μου Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ζητώ συγγνώμη που δεν βρισκόμουν στη θέση μου. Μου στήσατε να πάρω το λόγο. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια σειρά από ζητήματα συνδυαστικά, γιατί τέθηκαν εδώ μια σειρά από θέματα προ συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά ε, το ζήτημα των κεφαλαγορών και τη Unilever. Ε, στην τελευταία έκθεση αναφερόταν πω η Ένωση των Κεφαλαγορών θα μπορούσε να επιφέρει περισσότερη ε, σταθερότητα τελικά στον, στην οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εσεί είχατε τεθεί υπέρ αυτής της προσέγγισης ε, και ε, είχατε θεωρήσει και εσείς προβληματική την ε, πρόταση εξαγοράς από την πλευρά της της Unilever. Είχατε πει δηλαδή και εσείς ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και δεν θα πρέπει να προβούμε σε βιαστικές αποφάσεις σε ό,τι αφορά ειδικότερα ε, το ζήτημα των μετόχων. Ε, θα πρέπει δηλαδή να είμαστε πιο προσεκτικοί σε ό,τι αποφάσει ε, αποφάσεις που λαμβάνουμε. Και νομίζω πω και περιβολικά, για παράδειγμα, ζητήματα θα πρέπει να ληφθούν περισσότερο υπόψη και να προβλεφθούν συγκεκριμένε διατάξει σε ό,τι αφορά τι κεφαλαγορέ, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά εξαγορέ, συγχωνεύσει και ούτω καθεξή. Με άλλα λόγια, δεν θα πρέπει να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να αποφύγουμε επιχειρήσεις να ε, μην σκέφτονται αποκλειστικά και μόνο βραχυπρόθεσμα, να μην προσπαθούν και μόνο να επιτύχουν βραχυπρόθεσμο κέρδος. Κύριος Ντάσιμπλουμ. Ναι, ε, ο στόχος της Ένωσης είναι ακριβώς να αποδεσμεύσουμε περισσότερε πηγέ χρηματοδότηση για τι επιχειρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μην εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από τι τράπεζε και το χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ένας ε, ε, καπιταλισμός ε, που βασίζεται στους μετόχους θα πρέπει να είναι η προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε για το μέλλον. Ένα άκρατο τέτοιο καπιταλισμό. Νομίζω πως ε, εκείνο που θα πρέπει να επιτύχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μία προστασία σε περίπτωση, για παράδειγμα, εχθρικών εξαγορών ή συμπεριφορών των ε, μετόχων, όπου υπάρχει ακριβώ ε, κίνδυνο σε ό,τι αφορά το χαρακτήρα τη εν λόγω επιχείρηση ή όπου, για παράδειγμα, υπάρχουν ε, στρατηγική σημασία συμφέροντα τα οποία απειλούνται από μια τέτοια εξαγορά συγχώνευση, είτε κράτου μέλου είτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε μια σειρά από κράτη-μέλη ήδη υπάρχουν τέτοια νομικά πλαίσια ή επιτροπές οι οποίες εξετάζουν τέτοιου είδου εχθρικές εξαγορές και βρίσκουν τρόπους για να προστατεύσουν ακριβώ τι επιχειρήσει, τι εθνικέ αυτέ επιχειρήσει από εχθρικέ εξαγωγέ. Και νομίζω πω ναι, αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το εξετάσουμε από κοινού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού είμαστε μια αγορά. Και εμεί από την πλευρά μας θα προσφέραμε κάθε σχετική πρόταση από την πλευρά τη Επιτροπής. Στις κάτω χώρε, για παράδειγμα, εμεί εξετάζουμε αυτή την περίοδο περαιτέρω νομοθεσία για την προστασία των επιχειρήσεών μα, ομίλων μα όταν υπάρχουν τέτοιου είδου. Ε, απόπειρε εξαγορέ, στο πλαίσιο των οποίων θίγονται στρατηγική σημασία ε, συμφέροντα και οικονομικού χαρακτήρα, για παράδειγμα, συμφέροντα. Νομίζω, νομίζω πω πραγματικά εδώ θα μπορούσε να αξιοποιήσει το δικαίωμα πρωτοβουλία τη Επιτροπή και να κάνει μια πρόταση. Πολ, θε να δευτερολογήσει, ε, ένα μισή λεπτό ακόμα. Ναι, να συνεχίσω στα αγγλικά. Ναι, αναμένουμε με ενδιαφέρον μια τέτοια πρόταση από την Επιτροπή, αλλά μήπω θα μπορούσατε κι εσεί να θίξετε αυτό το ζήτημα είτε στο ECOFIN είτε στο Eurogroup. Γιατί διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο 100 χώρε, αλλά και άλλα κράτη-μέλη εξετάζουν νομοθετικέ λύσει και άλλου τρόπου για την προστασία των επιχειρήσεων του από εθνικέ εξαγωγέ. Ειδικότερα όταν πρόκειται για κρατικέ επιχειρήσει. Ε, υπάρχουν και κάποιε ανησυχίε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την Κίνα. Μήπω θα πρέπει να συζητηθούν αυτά τα ζητήματα από κοινού. Δεν θα πρέπει να το θέσετε κι εσεί, να αξιοποιήσετε δηλαδή το αξιωμά σα για να το θέσετε. Uh, Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη εξετάζει μια πιθανή πρόταση για το ζήτημα αυτό ενδεχομένως να βρίσκεται στη μερίσια διάταξη άλλων συμβουλίων και όχι στο ΕΚΟΦΗΝ Πάντω στι κάτω χώρε είναι το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων που ασχολείται με το ζήτημα αυτό. Εγώ έχω την προσωπική μου άποψη, αλλά δεν είμαι ο πλέον αρμόδιο για το ζήτημα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως ήδη επεξεργάζεται μια μελλοντική πρωτοβουλία για το ζήτημα αυτό. Και δυστυχώ, η πρωτοβουλία αυτή, λέει ο πρόεδρο, δεν θα είναι στην δική μα την Επιτροπή, αλλά θα εμφανιστεί στην Επιτροπή Εμπορίου. Επόμενος ομιλητής, Τόμ Φανέκαν Λάρε από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και εγώ θα μιλήσω Ολλανδικά. Έχουμε σήμερα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή το μερωτικό φυλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και λέει για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί περισσότερο το διορθωτικό σκέλο του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη, ιδίω για τι μακροοικονομικέ ανισορροπίε. Φαίνεται όμω ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κίνητρα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συμμορφωθούν ορισμένε χώρε. Εσεί έχετε μία μεγάλη εμπειρία ω πρόεδρο του Eurogroup. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει προκειμένου η διαδικασία αυτή να γίνει πραγματικά αποδοτική και αποτελεσματική η πολιτική βούληση από ό,τι φαίνεται από μόνη τη δεν φτάνει. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η πίεση από μοτίμους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του Eurogroup. Είπατε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσετε περισσότερο benchmarking. Έχει αυτό οδηγήσει σε άλλου τομεί σε καλύτερα αποτελέσματα στα κράτη-μέλη και Γέννη, θεωρείτε ότι το Eurogroup μπορεί να προωθήσει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τι δαθαπτικέ μεταρρυθμίσει. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Πιστεύω πραγματικά ότι έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες να αυξήσουμε την πίεση. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει προκειμένου να ασκήσει πίεση στα κράτη-μέλη, τόσο όσον αφορά τα σχέδια τα δημοσιονομικά και όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Πιστεύω επίση ότι πίεση ομοτήμων, όπως είπατε, μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο αρνητικά αλλά και εντελώ θετικά. Για παράδειγμα, στα πλαίσια του Eurogroup προσπαθήσαμε να δούμε πώ μπορούμε να μειώσουμε τη φορολογική επιβάρυνση τη εργασία, που είναι πάρα πολύ ψηλή στι χώρε Ευρωζώνη, πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Νομίζω ότι η Ιρλανδία βρίσκεται μόνο κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ και αυτή η φορολογική επιβάρυνση τη αγορά-εργασία δυσχεραίνει τη σωστή λειτουργία τη αγορά-εργασία και δεν μα στο να δημιουργήσουμε περισσότερε θέσει εργασία. Τα τελευταία χρόνια 5-6 χώρε έχουν κάνει φορολογικέ μεταρρυθμίσει, μειώντα τη φορολογική επιβάρυνση τη εργασία, ιδίω όσον αφορά το τμήμα εκείνων των, των ανθρώπων που έχουν χαμηλά εισοδήματα. Νομίζω λοιπόν ότι περισσότερε δραστηριοτικέ μεταρρυθμίσεις μπορούν να γίνουν σε όλε τι χώρε. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Τώρα από θεωρητική πλευρά θα ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνουν οι μεταρρυθμίσει τώρα που η οικονομία ανακάμπτει. Από πολιτική πλευρά όμω δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα από ό,τι φαίνεται. Από πολιτική πλευρά το αίσθημα αυτό της επίγουσας κατάστασης για περισσότερες μεταρρυθμίσεις κάπου χάνεται τελικά, καθώς απομακρυνόμαστε σιγά σιγά από την κρίση. Δυστυχώς. Δυστυχώς συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τόμ, έχεις ακόμα δύο λεπτά. Ένα ακόμα ερώτημα λοιπόν. Στην απάντησή σας στην Περβάνς Μπερές για το μέλλον της ε, ΟΝΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφερθήκατε σε μείγμα διαφορετικών σενάριων ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη εναλλακτική τελικά Αναφερθήκατε όμω στην πραγματική προστιθέμενη αξία που θα μπορούσαμε να είχαμε σε κάθε τομέα ξεχωριστά. Νομίζω το κάνατε αυτό. Αναφερθήκατε στην ε, δυνατότητα να επαναφέρουμε κάποιε αρμοδιότητε σε επίπεδο κρατών μελών. Πού πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, μπορείτε να μα δώσετε κάποια παραδείγματα. Απάντηση. Ναι, κοιτάξτε, έχω κάποιε παγιωμένε απόψει ω προ αυτό, αλλά ω πρόεδρο του Eurogroup καταλαβαίνετε ότι το ερώτημα αυτό και η απάντηση στο ερώτημα αυτό υπερβαίνει τελικά τι αρμοδιότητέ μου. Έχω διάφορε όμω ιδέε, τι οποίε δεν μπορώ να εκφράσω αυτή τη στιγμή ω πρόεδρο του Eurogroup. Σα ικανοποιεί η απάντηση αυτή, έχετε ακόμα ένα λεπτό. Δεν μπορείτε να είστε ικανοποιημένο προφανώ με αυτή την απάντηση. Ο τελευταίο ομιλητή από τι πολιτικέ ομάδε είναι ο κύριο Κώστα Μαυρίδη και μετά περνάμε στην διαδικασία uh, tongue. Uh, κύριε Ντάιζεμπλουμ, uh, πριν ένα μήνα είχαμε την έκθεση της Κομισιόν για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Και κοιτάζω στην έκθεση αυτή, η οποία διαπιστώνει ότι Βουλγαρία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Πορτογαλία και Κύπρος αντιμετωπίζουν excessive economic imbalances. Χθες και σήμερα τα δημοσιεύματα στον τύπο λένε ότι στο Eurogroup δόθηκαν εξηγήσει και σε πάρα πολλά από αυτά τα κράτη-μέλη που μόλις διάβασα, ενδεχομένως και όλα, να έδωσαν τέτοιες εξηγήσει που να ανατρέπουν τις διαπιστώσεις της Κομισιόν. Σας ρωτώ, πού είναι η πραγματικότητα, ποιος έχει την πραγματική εικόνα, η Κομισιόν ή το Eurogroup με βάση αυτά τα δημοσιεύματα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο είναι σχετικά με την Ελλάδα. Και συνάδελφοί μου εδώ και ιδιαίτερα ο κύριος Μπούλμαν αναφέρθηκε στο πρόβλημα που δημιουργείται από την έλλειψη σταθερότητας. Ε, στην ελληνική μυθολογία υπάρχει το τέρας της Λερναίας Ήδρας. Έκοβε ένα κεφάλι ο Ηρακλής, πετάγονταν δύο. Αναφερθήκατε στην αρχική σας εισήγηση για upfront structural measures, labor market reforms, που είναι collective labor bargaining. Όλα αυτά τα προβλήματα που μπαίνουν συνεχώς, ποιος τα επιβάλλει. Εσείς προσωπικά τα υιοθετείτε. Ευχαριστώ. Uh, uh, Τώρα στη συζήτηση που κάναμε στο Eurogroup συζητήσαμε την εφαρμογή των σχεδίων δημοσιονομικών ε, προγραμμάτων DBPs και εδώ η Επιτροπή και το αναγνωρίζει η δήλωση του Eurogroup το Δεκέμβριο η Επιτροπή λοιπόν τόνισε ότι 7 χώρες ήταν σε κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τα PPP αυτά και ότι θα έπρεπε να λάβουν συγκροματικά μέτρα. Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Άρα ίσως υπάρχει παρανόηση. Εσείς είπατε ε, υπερβολικές οικονομικές ανισορροπίες. Δεν συζητήσαμε αυτές στο Eurogroup χθες. Και οι χώρες που αναφέρατε δεν μας έδωσαν ε, εξηγήσει ε, που να απορρίπτουν τη θέση της Κομισιόν. Άρα η Κομισιόν έχει δίκιο. Δεύτερον, για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που είναι ακόμα αναγκαία στην Ελλάδα. Έχετε δίκιο. Αυτά είναι τα θέματα που εδώ και πολύ καιρό συζητάμε και έχουν ε, γίνει πράγματα. Έχει γίνει δημοσιονομική προσαρμογή. Αλλά βλέποντας σε βάθος χρόνου πρέπει να καταλάβουμε ότι οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από τις ε, διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις ήταν κυρίως δημοσιονομικού χαρακτήρα. Θα έλεγα από αυτή την πλευρά τα περισσότερα έχουν γίνει. Το βασικό όμως τώρα είναι να διατηρηθεί μια προσεκτική δημοσιονομική πολιτική, αλλά οι μεγάλη έκταση δημοσιονομικές προσαρμογές δεν χρειάζονται πλέον. Αυτό που χρειάζεται είναι περαιτέρω προσαρμογέ στην λειτουργία της αγορας εργασία, του, δημοσιο... του συνταξιωτικού συστήματο, την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματο κτλ. Αυτά πρέπει να γίνουν από οικονομική άποψη, ούτως ώστε αυτά τα συστήματα, αυτές οι αγορές να λειτουργήσουν καλύτερα για την Ελλάδα και για να διατηρηθεί η μακροπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές βεβαίως ε, θα χρειαστεί να συνοδευτούν από συμπληρωματικά βήματα. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι αν γίνουν κάποια επιπλέον βήματα για αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα μειωθεί η πίεση για περισσότερη λιτότητα. Και αυτή η έμφαση στην, στην λιτότητα νομίζω ότι είναι παρελθόν. Τώρα πρέπει να έχουμε ένα σαφώς διαφορετικό μήνυμα ότι πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα η οικονομία και ο δημόσιος τομέας για να γίνουν πιο βιώσιμα. Πρόεδρος, έχετε 15 δευτερόλεπτα. Ναι, λίγα λόγια. Πρώτον. Ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών πρότεινε τη δημιουργία της λεγόμενης κακής τράπεζας για τα «no performing loans. Έχετε άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Έληξε ο χρόνος όμως τώρα. Αυτό ήθελα να πω. Θα απαντήσετε. Πολύ σύντομα. Άλλοι τέσσερις έχουν το λόγο. Και πρέπει να τελειώνουμε. Κοιτάξτε, κάπως με προβλημάτισε η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, γιατί δεν ήταν σαφέ από πού από θα προέλθουν οι τεράστιοι αυτοί πόροι που θα προελθουν οι τεραστιοι αυτοι ποροι που χρειαζομαστε για να υλοποιηθεί η πρόταση αυτή. Και αν δημιουργηθεί μια νέα πολιτική bailout, μια νέα πρόταση bailout, εγώ θα ήμουν κατά. Και ουσιαστικά αυτό αντιβαίνει στα όσα λέμε αυτή τη στιγμή στα πλαίσια τη ε, οδηγία για την εξυγίανση των ε, τραπεζών. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο το bail-in και όχι το bail-out. Τέσσερι ακόμα μιλητέ θέλουν το λόγο, λέει ο Πρόεδρο. Από κοινού α ακούσουμε τι ερωτήσει αυτέ και θα ακούσουμε μετά τη συνολική απάντηση του κυρίου Ντάισελμπλουμ, γιατί πιέζει πάρα πολύ και ο χρόνο και έχουμε και την συνεδρίαση των συντονιστών αμέσω μετά. Ο κύριο Αργενόπλου έχει το λόγο. Για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ένα λεπτό ο καθένα από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ. Ε, σχετικά με το ελληνικό μνημόνιο και τι βέλτιστε ε, πρακτικέ. Κύριε Ντάισελμπλουμ, ε, στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι ξέρουν ότι με την ελληνική κυβέρνηση στην αξιολόγηση συμφωνείται για νέα μείωση μισθών. Ωστόσο και εσεί και η ελληνική κυβέρνηση για να εφησυχάσουν του εργαζόμενου και να του παραπλανήσουν μιλάνε για βέλτιστε πρακτικέ και ευρωπαϊκό κεκτημένο. Προχθές ο κύριο Μοσκοβισή, και έχω εδώ την απάντησή του, μίλησε για συλλογικέ συμβάσει εργασία που θα παίρνουν υπόψη τους την αντίστοιχη κακή προσθέτω οικονομική κατάσταση τη χώρα και τι διαρθρωτικέ αλλαγέ που οδήγησαν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Γαλλία και την Ιταλία που δεν έχουν μόνοι σε μέρου μισθών. Η κυρία Τάισεν σε ερώτηση δικιά μου σε γραπτή της απάντηση αναφέρει ότι οι συλλογικές συμβάσεις πρέπει να παρακολουθούν την παραγωγικότητα της εργασίας, δηλαδή να μειώνονται κάθε φορά που μια επιχείρηση επικαλείται μείωση παραγωγικότητας. Το ίδιο και το πρόβλημα εμπειρογνωμόνων. Τελικά, αυτό που εσείς ονομάζετε τελείωσα κύριε Πρόεδρε, φιλικό στι επενδύσεις σύστημα συλλογικών συμβάσεων και ευέλτιστες πρακτικές σημαίνει μειώσεις μισθών. bitte äh, auf eine Frage konzentrieren. Stephen Wolf ist next on my list. Stephen Wolf επόμενος και μετά ο Bernd Lücke. Ευχαριστώ. Ε, είπατε ότι βλέπετε κάποιες θετικές προοπτικές σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη της ε, ζουν στο ευρώ, αλλά εξφράζονται κάποιε ανησυχίε, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, τις, ε, τα κεφάλαια που εκραίουν από τι οικονομίε και το γεγονό ότι μόνο 5-6 χώρε ε, είναι εκείνε οι οποίε ε, τελικά τα αποκρίνουν τι υποχρεώσει του. Καθώς τώρα επίκειται και το Brexit και θα ξεκινήσει και επίσημα από την κυρία ε, Μέη η διαδικασία την ερχόμενη εβδομάδα και καθώς προετοιμάζετε και εσεί τι σχετικέ τις για του προπολογισμού στις 7 Μαου στο Συμβουλίο θα περιλάβετε ε, και κάποιε πτυχέ σε ό,τι αφορά την οικονομική πραγματικότητα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν όλε αυτέ οι χώρε εν ώψη ακριβώς και του Brexit. Γιατί όπω είπατε και εσεί δεν ακούσατε κάποιε ρεαλιστικέ προτάσει σε ό,τι αφορά τον περίπλοκο χαρακτήρα και τι δαπάνε που συνεπάγεται το Brexit. Οπότε υπάρχει κάποια τελικά ρεαλιστική εδώ εκτίμηση από πλευρά των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά το τι θα σημάνουν αυτέ οι δαπάνε κυρία Ντάσιμπλουμ, ε, στο ε, ε, σχόλια που κάνατε σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Ελλάδας, δεν αναφερθήκατε στο συζύγιο των 300 συναλλαγών, το οποίο ήταν θετικό για μια περίοδο, αλλά από το 2015 πλέον είναι ελληματικό. Άρα αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά ότι η Ελλάδα δεν είναι ανταγωνιστική τη σήμερα ημέρα. Εάν λοιπόν ε, τώρα ισχύουν οι αισιόδοξε ε, προβλέψει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ισχύουν και ότι δηλαδή υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, αυτό θα σημαίνει βέβαια ότι θα υπάρξει και αύξηση των εισαγωγών στην Ελλάδα, άρα περαιτέρω επιδείνωση αυτού του ίδιου τρέχουσων συναλλαγών. Πώ λοιπόν θεωρείτε εσεί πω θα καταφέρει η Ελλάδα να συνδυάσει τη βελτίωση δηλαδή αυτού του ισοζυγίου τρέχουσων συναλλαγών με την οικονομική ανάπτυξη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ντάσεμπλουν. Ε, ε, εκπροσωπώ μια από το Καταλωνία της ε, και είδα συμπατριώτε μου οι οποίοι εκνευρίστηκαν πολύ με τις δηλώσει που κάνατε στον τύπο σε ό,τι αφορά τις γυναίκες το ποτό. Ενδεχομένω, κάποια στιγμή στο μέλλον θα μπορούσατε να λέτε ότι ότι αντί ε, την επόμενη φορά μάλλον που θα στήσετε βοήθεια δεν θα πρέπει να επενδύετε σε έργα τα οποία δεν έχουν νόημα για παράδειγμα όπως ε, τρένα υψηλή ταχύτητα, τα οποία δεν έχουν επιβάτες όπως έργα δηλαδή όπως αυτά είδαμε και εμείς κατανοούμε κατά τα τελευταία ε, χρόνια. Ίσως λοιπόν την επόμενη φορά θα έχετε περισσότερα επιχειρήματα ή παραδείγματα να αναφέρετε ως προς το που δεν θα πρέπει να επενδύει η Ισπανία επιχειρήσεις για παράδειγμα οι οποίε ε, καλούνται να είναι αρμόδιε για τη διαχείριση τέτοιου είδου ε, τρένων τα οποία τελικά δεν λειτουργούν στην πράξη και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τα καθήκοντά σα και στο μέλλον κύριε Ντάση. Κύριος Ντάση μου έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Το πρώτο ζήτημα που αναφέρθηκε αφορούσε την Ελλάδα και σε ό,τι αφορά τι συλλογέ μας και το τι θα πρέπει τελικά να επιτρέπουμε ή όχι, αν δηλαδή στην ε, πράξη αυτό συνεπάγεται μείωση των μισθών. Και επειδή ακριβώ ε, η παραγωγικότητα λέτε, των επιχειρήσεων κατά επόμενα χρόνια στην Ελλάδα δεν θα αυξηθεί, θα συνεχίσει μειούμενη. Αλλά εγώ δεν συμφωνώ με αυτό ε, ότι δηλαδή θα συνεχίσει μια τέτοια μείωση τη παραγωγικότητα και δεν συμφωνώ με το ότι θα πρέπει να είναι συνδεδεμένε αυτέ οι ε, συλλογικέ διαπραγματεύσει με ε, την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά το ερώτημα των δαπανών που θα προκύψουν από το Brexit, πραγματικά ήταν πολύ κακή ιδέα το Brexit. Θα συνεπάγεται δαπάνε για όλου μα γιατί όσο πιο ισχυροί είναι και οι εμπορικοί δεσμοί τόσο πιο ε, υψηλό και το κόστο το οποίο θα κληθούμε να καταβάλουμε και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Στη δική μου χώρα, το CPP προείδησε σε κάποιες ε, σε κάποιους υπολογισμούς των δαπανών που θα προκύψουν ε, μακροπρόθεσμα ε, και πραγματικά είναι υψηλές αυτές οι δαπάνες. Οπότε μακροπρόθεσμα θα είναι υψηλότατες και θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Είναι κακή αυτή η ιδέα του Brexit, δεν ήταν δική μου ιδέα το Brexit και πραγματικά θα πρέπει να επιδείξουν όλες οι πλευρές ρεαλισμό. Όμω, βέβαια, ακούσαμε πολλά περισσότερα από την ευρωπαϊκή πλευρά μέχρι τώρα, ρεαλιστικά, από ό,τι από τη βρετανική. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημα, σε ό,τι αφορά τη δυνητική βελτίωση του ισοζυγίου τροχουσών συλλαγών της Ελλάδας. Ε, ουσιαστικά επιστρέφουμε στο ερώτημα του κατά πόσο μπορεί τελικά να καταστεί ισχυρότερη οικονομία η Ελλάδα. Μπορεί δηλαδή τελικά σε κάποια φάση η Ελλάδα να καταστεί ανταγωνιστική εντό τη ζώνη του ευρώ. Εγώ θεωρώ πω ναι, είναι δυνατό, αλλά θα χρειαστούν περαιτέρω ε, μεταρρυθμίσει, περισσότερε προσαρμογέ ε, στην οικονομία ε, σε ό,τι αφορά τι επενδύσει, την ανάκτηση τη εμπιστοσύνη των επενδυτών έτσι ώστε να επενδύσουν σε ευκαιρίε. Χρειάζεται σταθερό πολιτικό κλίμα, χρειάζεται μείωση της διαφθοράς, χρειάζεται δικαιοσύνη φορολογική, χρειάζεται προβλεψιμότητα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση ε, σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Όλα λοιπόν αυτά αποτελούν προ υποθέσεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου επιχειρησιακού κλίματος, αλλά χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά, σε αυτό συμφωνούμε. Και τέλος, σε ό,τι αφορά το τελευταίο ζήτημα που αναφέρθηκε σε σχέση με την Ισπανία, ναι, έλαβα υπόψη σας το σχόλιο αυτό, αλλά το δικό μου σχόλιο δεν αφορούσε κάποια συγκεκριμένη χώρα. Εγώ αναφέρθηκα στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση τη Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο πρόεδρο, τον κύριο Ντάισεμπλουμ για την παρουσία του σήμερα εδώ και τις απαντήσεις που έδωσε σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν. Πραγματικά ποικίλα ερωτήματα τέθηκαν σήμερα το απόγευμα. Υπό το σημείο 4 της ημέρας σας διάταξης δεν έχω τίποτα από τα διάφορα. Ε, αύριο λοιπόν το πρωί η συνεδρίασή μας η κανονική συνεχίζεται στις 9 το πρωί, οπότε ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση. Όσοι λοιπόν δεν είναι συντονιστές, τους παρακαλώ να αποχωρήσουν άμεσα, ώστε να συνεχίσουμε απευθείας με τη συνεδρίαση των συντονιστών.